Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Είστε παρακαλώ. Starten, dann... Ξεκινάμε. Και θα ήθελα, αν δεν έχει κανείς αντίρρηση για την ημερήσια διάταξη, να θεωρήσω πως εγκρίνεται. δεν βλέπω καμία αντίρρηση, οπότε εγκρίνεται όσον αφορά τη ερμηνεία. Εκτός από τα ιστονικά και τα μαλτέζικα και τα κροατικά έχουμε όλες τις γλώσσες. Έχουμε ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας. Καλωσορίζω τον Μακ Ντεμσμέκερ. Είναι και παρόν. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Και αντικαθιστά την συνάδελφο την Φρίντα Βρέπουλς. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών. Τον κύριο Νικολάη Άστρουπ, ε, Νορβηγός βουλευτής. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση ε, Μετάφρασης από το Λουξεμβούργο, 16 εκπαιδευόμενοι, δεν τους βλέπω εγώ, κάπου εδώ θα είναι. Τέταρτη ανακοίνωση, έχουμε εργαστήριο της ομάδας εργασίας ε, για την υγεία, για τα ε, ιατρικά προϊόντα προωθημένης θεραπείας και την εφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτό στις 20 Φεβρουαρίου από 1 μέχρι 2 και 40 στην Α3Ε3 και το εργαστήριο για τα βιοκαύσιμα και αυτό στις 20 Φεβρουαρίου 3 με 6 στην α 3 Α3Ε2 και υπάρχει και μια συζήτηση για τις ιατρικές συσκευές και ε, συσκευές in vitro 26 Φεβρουαρίου από τις 12.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα στην 1G2 την αίθουσα του κτηρίου ASP. Μετά περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης οχήματα και πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι του διοξιδίου του άνθρακα από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κράμερ, τον οποίο ε, δίνω αμέσως το λόγο για να κάνει μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Ε, Jetzt, jetzt geht's. Ja. Äh, gut bekannt sein, Πρέπει νομίζω να τα ξέρετε τα θέματα, γιατί πριν από δύο χρόνια τα είχαμε ξανασυζητήσει, ήταν επίμαχο θέμα, τότε το διοξείδιο του άνθρακα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Η συζήτηση την οποία είχαμε τότε αφορούσε τους στόχους για το 2020. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση και θα θυμάστε τα 147 γραμμάρια, τα περίφημα για το μέσο όρο του συνόλου του στόλου. Θυμάστε πως στάσαμε σε αυτό το νούμερο. Η Κομισιόν τώρα είχε την αποστολή μέχρι πέρσι να ε, εξακριβώσει την ε, σκοπιμότητα και τις ε, λεπτομέρειες εφαρμογής του στόχου αυτού. Το έκανε λοιπόν, εμείς πρέπει τώρα να απαντήσουμε. Δεν ε, υπήρξαν νέε εξελίξεις, δεν προσαρμόστηκαν τα πράγματα, αλλά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση για το ερώτημα αν αυτός ο στόχος ε, είναι αρκετά φιλόδοξος για το 2020, πως πρέπει να βελτιωθεί, αν υπάρχουν νέες πληροφορίες, νέα επιχειρήματα για να αλλάξει κάτι και εγώ στους τελευταίους μήνες και εβδομάδες άκουσα πάρα πολλά επιχειρήματα από πολλές πλευρές και θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, που ήταν και στην ακρόαση, ακούστηκαν πάρα πολλά επιχειρήματα. Στο σχέδιο έκθεση λοιπόν που έχετε τώρα μπροστά σας ε, αποφάσισα ξεκάθαρα να μην αλλάξουμε τίποτα στο στόχο του 2020. Το βασικό επιχείρημα είναι πως πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία στους ε, βραχυπρόσιμους στόχους μας ε, και δεν μπορούμε τώρα 7 χρόνια πριν το 2020 ε, και λιγότερο από 2 χρόνια από όταν θέσαμε το νούμερο αυτό να το αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς της αυτοκινητοβιομηχανίας για να καταλάβει πως ο κύκλος παραγωγής ενός φορτηγού είναι πολύ μεγαλύτερος από τον γιοταχή. Οπότε ακριβώς τα ελαφρά αυτά φορτηγά και οχήματα και είναι ε, τώρα στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής θα είναι στους δρόμους το 2020 οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφάλεια του σχεδιασμού και βεβαίως γνωρίζω την συζήτηση αυτή. Έχω δει μελέτες που λένε πως ε, μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Έχω δει μελέτες που λένε πως με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες και τις προβλέψιμες ε, ε, δυνατότητες ίσως να μην ε, είναι τεχνολογικά εφικτά τα 147 γραμμάρια. Οπότε αυτό βεβαίως εξαρτάται και από την κάθε μελέτη που διαβάζει κανείς, αλλά δείχνει πως η, κατάσταση μας συγχωρείτε είναι ακόμα αβέβαιοι. Και βεβαίω ε, είναι ευρύτατη αυτή η αγορά με διάφορες τεχνικές προδιαγραφές, γι' αυτό εγώ θα πρότεινα να μην πειράξουμε το στόχο του 2020 και εγώ θα υποβάλω μια μελέτη ε, τις επόμενες ε, ε, εβδομάδες που αμφισβητεί ακόμα και τα 147, τα οποία ίσως είναι υπερβολικά φιλόδοξα. Δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά τη συζήτηση για τα γεωταχή. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό ανεξάρτητα από τον κύκλο δοκιμών με τον οποίο διαπιστώνεται. Γι' αυτό πρέπει να πούμε πως όταν αποφασιστεί και οριστεί και μπορεί να εφαρμοστεί ένας νέος κύκλος δοκιμών και δεν είναι αυτό πολιτικό το ζήτημα, είναι μαθηματικό γιατί όταν αλλάζουν βεβαίως οι παράμετροι αλλάζουν ε, ε μεταβλητές ε, το αν είναι αναμένο το air condition, ε, η ταχύτητα του οχήματος κτλ. Και εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει κάποια ασφαλεία σχεδιασμού. Οπότε η πρότασή μου είναι όταν υπάρξει ένας νέος ε, κύκλος δοκιμών να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό, να δούμε. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση πω οι συζητήσει στον ΟΗΕ είναι προχωρημένε, αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει για την περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο να έχουμε αξιόπιστα νούμερα στην περίπτωση που θα έχουμε τον παλαιό κύκλο δοκιμών. Ε, η Κομισιόν έχει δώσει μια ημερομηνία στόχο για μετά το 2020, η οποία πήγε πιο πίσω. Εγώ δεν θέλω να δω το 2018, δεν θα ήθελα το 2018. Το ένα είναι βεβαίως ο κύκλος των δοκιμών αλλά το άλλο είναι βεβαίως το τι θα γίνει μετά το 2020, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ε, υπάρχουν νέες τεχνολογίες, ε, υβριδικά, ηλεκτρικά, αυτοκίνητα, αέριο, πολλές εναλλακτικέ και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς και πότε και σε ποιο βαθμό θα ε, είναι διαθέσιμα στην αγορά. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο για να ξέρουμε τι θα γίνει μετά το 2020. Στην έκθεσή μου έγραψα κάτι το οποίο δεν έκανε η Κομισιόν δύο επιχειρήματα τα λεγόμενα super credits, ότι υπολογίζονται δηλαδή πολλές φορές ε, τα οχήματα στον υπολογισμό των εκπομπών, κάτι το οποίο γίνεται για τα γεωτοχεία, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται για τα ελαφρά φορτηγά, ειδικά σε αυτόν τον τομέα, όταν μιλάμε δηλαδή για αστικές περιοχές, εκεί πέρα πέρα από τα γιοταχή και σε αντίθεση με τα γιοταχή υπάρχει νομίζω πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ηλεκτρικής ε, κίνησης και τα super credits αυτά θα μπορούσαν να είναι ένα κίνητρο για να αλλάξουμε τεχνολογία χωρίς να επιβαρυνθεί και ο φορολογούμενος. Και αυτό με το επιχείρημα που λέει πάντα η Κομισιόν. Πρέπει να μην εξαρτώμαστε πλέον από τα ορυκτά καύσιμα, να περιοριστεί αυτή η εξάρτηση και να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Και ακριβώ ε, στα ελαφρά φορτηγά υπάρχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες. Να μιλάμε για στόλους ε, εταιριών που κάνουν ε, παραδόσεις κτλ. Εκεί πέρα οι νέες τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα άλμα προς τα εμπρός. Τελευταίο, έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή, μια περιβαλλοντική ένωση, την οποία διάβασα και είχε υπογραφεί και από κάποιες εταιρείε. Ήταν ένα ξεκάθαρο lobbying ε, αναξιόπιστο, γιατί ε, μια μελέτη κατέδειξε πως ε, δεν συζητάει κανείς αυτή την απέτηση την οποία είχαν για αυστηροποίηση Γι' αυτό ε, δεν ε, το συζητάω καν ε, αυτό το οποίο αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή και ζητώ όταν σας κάνουν lobbying ε, να κοιτάτε λίγο και την αξιοπιστία αυτών που ζητάνε τα διάφορα πράγματα και των πληροφοριών επίσης. Εγώ δυστυχώς ε, είμαι στόχος διαφόρων απόψεων που με φτάνουν από διάφορες ομάδες συμφερόντων. Αυτά για την έκθεση. Αναμένω βεβαίω τη συζήτηση, τις διαπραγματεύσει και ελπίζω να ολοκληρώσουμε σχετικά σύντομα γιατί δεν είναι αυτή τώρα μια μεγάλη συζήτηση αρχών. Το θέμα είναι να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Γκροστέτ, η οποία εκπροσωπείται από τον κύριο Ταρέλα. Εκπροσωπεί τον κύριο Ταταρέλα. Ευχαριστώ. Λαμβάνω το λόγο εξ του κυρίου Ταταρέλα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα. Γενικά συμφωνεί με τις προτάσεις που, έχει διατυπωθεί, που έχουν διατυπωθεί στην έκθεση του κυρίου Κράμερ, αλλά ο κύριος Ταταρέλα διατηρεί κάποιες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά το στόχο των 147 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακος ανά χιλιόμετρο θεωρώντας ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος αυτός ο στόχος, υπερβολικά φιλόδοξος, σε μια φάση οικονομικής κρίσης, θεωρεί λοιπόν ότι θα ήταν πιο πρέπον να μην επιβάλλουμε περαιτέρω ρυθμιστικές, ε, ρυθμιστικά άχθη στους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Θεωρεί ότι τα πριμ είναι θετικά σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προώθησης της τεχνολογικής αλλαγής και σαν κίνητρα για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπο. Επίσης είναι και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει και με αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων αυτού του κανονισμού χωρίς του κανονισμού 2011 χωρίς να επιβάλλει πρόσθετα βάρη στους φορολογούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση αυτών των κινήτρων και των πριμ επιτρέπει να προωθήσουμε κάθε είδους εναλλακτικές μορφές ε, προώθησης των οχημάτων και μηχανοκίνησής τους. Επομένως θα πρέπει να παραταθεί η ισχύ αυτού του κανονισμού μέχρι το 2018 όπως προβλεπόταν στην ψηφοφορία που είναι αυτού του κανονισμού του 2011. Αυτά θέλω να μεταφέρω λοιπόν εξ του κυρίου Ταταρέλα και σας ε, αναφέρω θα ζητήσω και πάλι το λόγο αλλά θα μιλήσω προσωπικά αργότερα στη συζήτηση αν αυτό είναι δυνατό. Ευχαριστώ λέει και η Μαρία Ταοσκότ για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Κράμερ αποτελεί και μία μορφή σφαγής της πρότασης της Κομισιόν και νομίζω ότι ο κύριος Κράμερ προχώρησε υπερβολικά μακριά. Αναφέρεται στους ε, στόχους του 2020, τα 147 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος. όλη αυτή η στόχοι είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μείωση των εκπομπών, αλλά ο τομέας των μεταφορών είναι ένας τομέας ο οποίος απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα για να παραμείνουμε πιστοί στον στόχο αυτό και να συνεχίσουμε να θεσπίζουμε φιλόδοξους στόχους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πρόταση της Κομισιόν. Όταν πρόκειται συγκεκριμένα για, τα, για τις απαιτήσει που γίνονται για τα οχήματα και ιδίως τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο φιλοδοξίας. Όπως ξέρετε, αυτό είναι μια παρακινδυνευμένη διαδικασία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη απόκληση των τεχνικών προδιαγραφών μεταξύ διαφορετικών είδων οχημάτων. Αυτό οδηγεί σε περιπλοκές. Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα μπορούν, θα μπορούν να απολούνται πολύ πιο εύκολα και αυτό θα έχει συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα ίδια αυτά οχημάτων τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και οι στόχοι μας να έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το στόχο. Αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα όπως θέλαμε. Σε ό,τι αφορά τους μακρό, μακρόπνους στόχους, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι, προσπαθώντας να μην δημιουργήσουμε στρεβλώσεις και μεγάλες αποκλήσεις για τη μεταχείριση των διαφορετικών ειδών οχημάτων. Πρέπει ο στόχος μας είναι να τροποποιήσουμε και την αντιμετώπιση των καταναλωτών και τις, ε, τις επιλογές σε επίπεδο αγορών των καταναλωτών για αυτά τα αυτοκίνητα. Για τις ε, εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών έχουν ποταθεί εδώ νέες εξαιρέσεις επί τη βάση του όγκου των οχημάτων αυτών και εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα κίνητρο για οποιονδήποτε. Γι' αυτό έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό για το συγκεκριμένο αυτό θέμα των εξαιρέσεων. Και σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα super prim, τα, τα, τις επιδοτήσεις αυτές, νομίζω ότι τον, το μέλλον αυτών ε, επιδοτήσεων θα πρέπει να εξαρτάται από το επίπεδο το οποίο θα επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών. Νομίζω ότι αυτές οι μορφές υπερπριμ μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο, μπορούν να αρρωγήσουν την διαδικασία για την ε, θέσπιση αυτού του καθεστώτος και την λειτουργία του. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις λεπτομέρειες και τώρα, σε σχέση με τα όρια ταχύτητας που θα επιβληθούν στα οχήματα αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και στο παρελθόν. Στην αρχή τη συζήτηση αυτή που. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Ο Κάρλ Σλούτερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριο Σλούτερ. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους. Οι στόχοι είναι σε επίπεδο κλιματολογικό. Προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς βοηθώντας τα κράτη-μέλη. Αν διευρύνουμε τις φιλοδοξίες μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε θα έχουμε μικρότερο κόστος εφαρμογής. Στην ουσία λοιπόν εξοικονομούμε τα χρήματα των καταναλωτών, των φορολογουμένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχοθετώντας ψηλότερα από ότι τα 175 τα οποία είχαν ε, βασιστεί σε ένα λανθασμένο υπολογισμό σε σχέση με το τι παράγουν τα σημερινά οχήματα. Πρέπει να μειωθούν λοιπόν τα επίπεδα αυτά τα ανώτατα γιατί είχαμε κάνει λάθος τον υπολογισμό τους. Αν δεν φανούμε πιο αυστηροί εδώ, τότε την εξοικονόμηση σε διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να την κάνουμε αλλού. Γι' αυτό θα κοστίσει. Πώς θα εξηγήσετε λοιπόν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που εξυπηρετούνται από ξυλουργού, ε, ξυλουργούς, από υδραυλικούς. Θα τους πούμε ότι εμείς θα υπερψηφίσουμε ένα κανονισμό ο οποίος θα αυξήσει το καθαρό κόστος εκμετάλλευσης των οχημάτων τους κατά 4-5 χιλιάδες ευρώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αυτοκινήτων τους. Όχι, αυτό είναι αδικαιολόγητο. Πρέπει να εξοικονομήσουμε τα χρήματα αυτά. Και το να λέμε στις επιχειρήσεις ότι ας παράγεται περισσότερη διοξίδιο του άνθρακα για να εξοικονομήσετε χρήματα, αυτό είναι ψευδέστηση. Κοιτάξτε, το 2020 σε ποιους θα πολλάμε τέτοια οχήματα. Ε, οι Κινέζοι και οι Ινδοί θα αγοράζουν ε, βενζινοβόρα αυτοκίνητα από εμά, όχι βέβαια. Κοιτάξτε, θα πρέπει να εξηγήσουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι το μέλλον βρίσκεται στην εξοικονόμηση χρημάτων, στην εξοικονόμηση μόλυνσης, στην εξοικονόμηση εκπομπών. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση το να μείνουμε στα σημερινά επίπεδα δεν θα βοηθήσει. Σχετικά με την προσθήκη των super credits, αυτό είναι απαράδεκτο γιατί οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει είναι ευκόλως επιτεύξιμοι. Οπότε θα τους καταστήσουμε πιο εύκολους. Αυτό θα είναι πραγματικά άχρηστο. Πού θα είναι η ευρωπαϊκή καινοτομία. Όλοι μιλάτε για καινοτομία. Αλλά εδώ λέμε εντάξει ας μην καινοτομήσουμε και πολύ, ας κρατήσουμε τα παλαιού τύπου και τεχνολογίας οχήματα. Αυτό δεν είναι το μέλλον θα συμφωνήσω με την Οσκοκό ότι οι περιοριστές ταχύτητας, οι κόφτες ταχύτητας είναι μια καλή ιδέα. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι νέες μορφές ελέγχου των αυτοκινήτων. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε απάτες σε σχέση μόνο με το αλογίσιο κρέας, έχουμε απάτες σε σχέση με ε, τις εκπομπές καυσαερίων, διότι τα τεστ στα οποία υποβάλλονται τα οχήματα είναι γεμάτα ε, κόλπα και κομπίνες. Λοιπόν, να σταματήσουμε να εξαπατούμε και να λέμε ψέματα στους φορολογουμένους. Ας δημιουργήσουμε ένα κύκλο ελέγχου των εκπομπών των αυτοκινήτων που να είναι αξιόπιστος και έτσι οι καταναλωτές να ξέρουν τι αγοράζουν και αν θέλουν να αγοράζουν βενζινοβόρα και να πληρώνουν φόρους σας το κάνουν. Αλλά αν θέλουν να είναι ευφυείς και να διασώζουν το περιβάλλον να γνωρίζουν ακριβώς τι εκπέμπουν τα οχήματα που αγοράζουν. Λοιπόν, για την οικονομία, για την καινοτομία, για το μέλλον απαιτούνται αυστηρότερα επίπεδα και δεν χρειάζονται τα super credits. Νομίζω ότι οι περιοριστές ταχύτητας είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Μπορεί να αυξήσει επίσης ε, οι κόφτες. Πρέπει να ε, θα περιορίσει και τα ατυχήματα στις οδικές ε, μετακινήσεις. Εντάξει, αυτό θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν. Ο Μάρτιν, ο Μάρτιν Κάλανεν δεν είναι παρόν. Είναι μαζί με τον κύριο Φων Ερχόμαστε στους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Λεπάζω έχει το λόγο τώρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα οποία ελέγχθηκαν μόλις, υπεθυμίζοντας ότι η στόχη της Κομισιόν το 2009 ήταν τα 136 γραμμάρια. Αν εφαρμόσουμε στα επαγγελματικά οχήματα το επίπεδο που θέλουμε για τα ελαφρά αυτοκίνητα θα ήταν, ήταν 136 γραμμάρια, επομένω τα 147 δεν είναι φιλόδοξα, είναι αντίθετα πολύ υψηλό επίπεδο και δεν μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας έναντι της κλιματικής αλλαγής, ούτε μας επιτρέπουν να φτάσουμε και φιλόδοξους στόχους σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής. Σε πολλές από τις χώρες μας η αυτοκίνητο βιομηχανία περνάει μεγάλες δυσκολίες. και μόνο με το να τους παρακινήσουμε και να τους πιέσουμε να προχωρήσουν προς αυτοκίνητα του 21ου αιώνα, αυτοκίνητα πιο ελαφρά, με μικρότερη κατανάλωση και λιγότερες εκπομπές, μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το βιομηχανικό αυτό τομέα της βιομηχανιας Έχουμε λοιπόν ένα συμφέρον το οποίο είναι και οικονομικό και βιομηχανικού χαρακτήρα, να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε σαφείς στόχους και να του εφαρμόσουμε το ταχύτερο το Χρειάζεται ένα βιομηχανικό κλάδο να έχει μια σαφή ορατότητα. Το να μην δώσουμε τώρα ορατότητα σε αυτό το τομέα, περιμένοντα το 2018, γιατί όχι το 2020, το 2025, όπω λέει και η κολοκυθιά, όλα αυτά θα δυσκολέψουν και θα κάνουν αδύνατη την πραγματική εξέλιξη στον τομέα της βιομηχανίας γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική προβλεψιμότητα για τις βιομηχανίες για να μπορέσουν να σχεδιάσουν την επόμενη γενιά αυτοκινήτων. Για όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από ό,τι προτείνεται αυτή τη στιγμή και από την Κομισιόν και από την εκθέση του κ. Κράμερ, παραμένοντας φυσικά ρεαλιστές, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική οικονομική συγκυρία για τα super credits, τα υπερπριμ. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα επεκτείνουμε περισσότερα, γιατί σε τελική ανάλυση τα επομίζεται ο Ευρωπαίος φορολογούμενος σε ένα δυσμενές πλαίσιο οικονομικό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει επομένως να ζητήσουμε την επέκταση αυτού του μέτρου. Για τους κύκλους δοκιμασίας θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις εκπομπές για ένα τομέα ο οποίος στην περίοδο αναφοράς αύξησε κατά 25% αυτές τις εκπομπές. Πρέπει να έχουμε πραγματικές δοκιμασίες και όταν βλέπουμε την κατανάλωση και τις εκπομπές διοξίδιου του άνθρακος, αυτές θα πρέπει να είναι σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε ιδανικές και εξωπραγματικές συνθήκες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν την διαφάνεια και το γενικό συμφέρον για τις δοκιμασίες αυτές. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Αλέπας. Εγώ συμφωνώ ιδιαίτερα με τον κύριο Κράμερ. όταν τονίστηκε ότι είναι όταν τόνισε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια μακροχρόνια σταθερότητα και ασφάλεια, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχει συμπεριλάβει και στην έκθεσή του. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μέχρι το 2018 δεν μπορούμε να χρονοτριβήσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο των 147 γραμμαρίων. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφυσβήτηση από κανένα. Όταν όμως είναι ανεδαφικός αυτός ο στόχος, μπορώ να δείξω και εγώ επιστολές που έχω λάβει και να πω στον κύριο Κράμερ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο στόχος γιατί αυτό θα είναι το τέλος του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Αν θυμάστε την οδηγία για, τα, για τις εκπομπές, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε πει ότι τέρμα δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε πια αυτοκίνητα. Και αντίθετα έγινε δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι του 2015 το 2012 παρά τις διαμαρτυρίες των ε, μεγάλων εταιριών. Μπορώ λοιπόν να σας ε, συγχαρώ για την κατεύθυνσή σας Πάντα διαμαρτύρονται οι εταιρείε όταν τίθενται οι προδιαγραφέ και μετά όταν εφαρμόζονται λένε τι ωραία έχουμε αυτά τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο και κάθε χρόνο χρειαζόμαστε λιγότερα καύσιμα για τα δυνατά και γρήγορα αυτοκίνητά μας. Είναι απαραίτητο όμως να έχουμε και στο μυαλό μας ένα ορίζοντα ο οποίος να είναι και επέκεινο του 2020 και όχι μονάχα ως το 2018 και θα πρέπει να παρακινήσουμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για τον κύκλο δοκιμασιών δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα, μεγαλύτερη κομπίνα από αυτό τον κύκλο δοκιμασιών. Φτάνουν να βάζουν λευκοπλάστη στις πόρτες οι κατασκευαστές για να μειώνουν την αντίσταση στον αέρα. Κάνουν τέτοια κόλπα. Δεν πρέπει εμείς να δεχόμαστε όλες αυτές τις διαδικασίες, όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν οι βιομηχανίες για να μειώσουν τις τιμές που προκύπτουν από τις δοκιμασίες. Και επίσης το δεύτερο ψέμα είναι ότι αυτός ο κύκλος αντιπροσωπεύει μια ε, λογική κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε λοιπόν επιτύχει πολλά πράγματα με αυτές τις δοκιμασίες. Πρέπει εμείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσουμε ότι λέμε την αλήθεια στους καταναλωτές μας και όταν θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο να ξέρουν ότι η δοκιμασία αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ε, ε, συνθήκες και όχι όταν τις κάνουν σε πραγματικές συνθήκες να βγαίνουν διπλάσιες αυτές οι τιμές από αυτά που έχει ο κύκλος δοκιμασίας. Δεν πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτά τα τεχνάσματα και τα οποία ευνοούν ίσως την αυτοκινητοβιομηχανία και θα τα γνωρίζω και ως Γερμανός, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πιο ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να είναι εφικτές οι διαδικασίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Εγώ είμαι φίλος των super credits, των, ε, πριν αυτόν. Εγώ θέλω να ζητήσω να υπάρξει και μια οροφή για αυτά τα, για αυτά τα πριμ. Να μην είναι ανοιχτή η χρησιμοποίησή τους και η επέκτασή τους. Εάν πρόκειται μονάχα για δύο ή τρία γραμμάρια μείωση της, ε, των εκπομπών, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε υπερπριμ τα οποία θα δίδονται στις ε, βιομηχανίες. Επομένως, αυτό δεν είναι επαρκές. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ε, πω, ας το δούμε το θέμα κανονικά. Εγώ δεν θέλω να τροποποιήσουμε το στόχο του 2020, αλλά δεν πρέπει να φέρουμε τον εαυτό μας σε πιο δύσκολη κατάσταση. Με τις ρυθμίσεις που κάνουμε τα αυτοκίνητα γίνονται πιο ακριβά. Είδαμε στο παρελθόν τα αυτοκίνητα να είναι 2.000 3.000 ευρώ πιο ακριβά, αλλά με τη μικρότερη κατανάλωση μέσα σε τρία χρόνια είχαν καταφέρει να αποσβέσουν οι ιδιοκτήτες τους αυτό το πρόσθετο κόστος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι σε ό,τι αφορά τους στόχους εξοικονόμησης και να καταφέρουμε να πείσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία να πουλάει αυτοκίνητα που έχουν πιο αποδοτικούς κινητήρες. Χρειάζεται κάποιο μέτρο. Και ο τρόπος με τον οποίο διενεργεί η αυτοκινητοβιομηχανία της συζήτησης αυτή είναι λαθασμένος. Μετά από τον ομιλία του Καλ Χάιντς Φλόρενς ε, αναμένω ήδη με αγωνία τις ε, ψηφοφορίες και πόσα από αυτά θα τηρήσει. Γεγονός είναι Καλ Χάιντς πως η αυτοκινητομηχανία πρέπει να βελτιωθεί κατά πολύ. Έχουμε τον οδικό χάρτη 2050 όπου είναι ξεκάθαρο πως οι μεταφορές πρέπει να συνεισφέρουν κατά 60% σε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή χρειάζονται θαραλέα βήματα. Δεν το συζητάω. Και θεωρώ πως ε, έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου υπάρχει τεχνολογικός μετασχηματισμός. Ε, τώρα θα προκύψουν νέοι κινητήρες, ε, νέες τεχνολογίες και έχουμε πολλές δυνατότητες. Και το Κοινοβούλιο μας, η Επιτροπή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Και αυτό το λέω γιατί εγώ είμαι υπέρ του στόχου να διατυπώσουμε ένα στόχο τώρα για το 2025. Το 2008 θέσαμε ένα στόχο για το 2020, δηλαδή 12 χρόνια στο μέλλον. Εντάξει, και τότε για να συζητήσει, αλλά είναι εφικτό. Τώρα είμαστε στο 2013 αν διατυπώσουμε ένα στόχο για 12 χρόνια στο μέλλον, είμαστε το 2025. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον πως ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το έχουμε ήδη κάνει μια φορά, πρέπει να το ξανακάνουμε. Για να ξέρει και η βιομηχανία που πάμε. Και θα είναι σε θέση να εφαρμόσει στην πράξη την τεχνογνωσία της τα αυτοκίνητα δεν είναι μόνο να δείχνουμε τα πρωτότυπα στα σαλόνια αυτοκινήτου, αλλά να τα φτιάχνουμε κιόλα. Και υπάρχει βεβαίω ένα πρόβλημα, το ότι είναι ακριβότερα αυτά τα αυτοκίνητα, αισθητά ακριβότερα. Και ε, πρέπει να μειωθεί το κόστος και μειώνται και τα κέρδη. Και οι καταναλωτές βεβαίως δεν ξέρουμε αν είναι διατεθειμένοι να τα αγοράσουν. Και το ερώτημα τίθεται πώς πρέπει να υπάρξει κάποιο κίνητρο για τη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες. Αυτό το λέμε λοιπόν υπερπιστώσεις. Εγώ δεν είμαι κατά των κινήτρων επί της αρχής, γιατί τα έχουμε δει αυτά τα αυτοκίνητα, υπάρχουν ως πρωτότυπα αλλά δεν κατασκευάζονται. Χρειάζεται λοιπόν ένα μέσο για να περάσουν στην παραγωγή και στην αγορά. Και όταν λέγεται credits, η κυρία Κορυλαπάς δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει ο φορολογούμενος ε, κάποια επιδότηση. Είναι ένας τρόπος έτσι, υπολογισμού. Οπότε φέτος ή του χρόνου το αργότερο πρέπει να ορίσουμε ένα στόχο το 2025 για τα super credits επίσημη υπέρ. Πρέπει βεβαίως να δούμε ε, πόσο θα είναι. Μην είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα κίνητρο. Επίσης, βλέπω πως γίνονται διάφορα με τον κύκλο δοκιμών. Δεν μπορώ να φανταστώ πως χρειάζεται τόσος χρόνος για να φτιάξουμε ένα σωστό και διάφανο κύκλο δοκιμών. Εγώ προτιμώ έναν καλύτερο κύκλο δοκιμών, γιατί, το οποίο θα έχουμε και ως μέτρο. Γιατί ο τωρινός είναι απλά απάτης βάρος του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Θα μιλήσω προσωπικά εδώ, όχι σαν εκπρόσωπος ομάδας. Πιστεύω ότι η έκθεση του κ. Κράμερ είναι μια θετική έκθεση. Και το όριο των 147 δεν θα πρέπει να αλλάξει. Είναι αρκετά φιλόδοξο στόχος. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά σήμερα και ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση αγοράζονται περισσότερα μεταχειρισμένα τέτοια οχήματα παρά νέα οχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε τα πράγματα λίγο πιο σχετικά παρακαλώ. Και όταν ακούω τον συνάδελφο Φλόρενς που λέει κοιτάξτε αν υπάρξουν αυξήσεις αυτό το 2-3 χιλιάδες επιπλέον ευρώ για τη ζωή ενός ελαφρού μεταφορικού οχήματος. Ε, κοιτάξτε 2-3 χιλιάδες ευρώ είναι απίστευτα υψηλό ποσό, ανυπόφορε υψηλό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί εδώ, να δούμε τι ακριβώς θέλουμε. Όταν θέλουμε να επιβάλλουμε κανόνες πιο δεσμευτικούς και πιο αυστηρούς στις αυτοκινητοβιομηχανίες για τα οχήματα αυτά, τότε θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τις ε, εκπομπές καυσαερίων. Σχετικά τώρα με τα, με αυτά είναι τμήμα της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και για το ιδιωτικά αυτοκίνητα, για ιοταχή οχήματα. Αλλά δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση για τα εμπορικής χρήσεως. Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα πρίμα αυτά είναι ένα μέσο το οποίο θα επιτρέψει να τεθεί στην αγορά και σε λειτουργία ένα σύστημα με νέα αυτοκίνητα νέου τύπου με χαμηλά επίπεδα εκπομπών και χωρίς να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Θέλει επίσης να φτάσουμε στο 165 για να συμπεριλάβουμε και τα μεγαλύτερου μεγέθους οχήματα και αυτό δεν είναι λάθος. Θα πρέπει εγώ να φτάσουμε στα 50 γραμμάρια γιατί κάποιοι κατασκευαστές καταφέρνουν ήδη στο όριο αυτό να φτάνουν γιατί ίσως τα 75 να μην βοηθήσουν α, ιδιαίτερα στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Κοιτάξτε, αυτά που συζητάμε τα είχαμε αποφασίσει το 11 και τώρα στο 13 θέλουμε να τα αμφισβητήσουμε όλα. Ας φανούμε λίγο ρεαλιστές, κοιτάξτε ποια είναι η κανονική χρήση κρίση και ποιες είναι οι αγοραστικές ικανότητες των χρηστών αυτών των οχημάτων. Ωραία. Έχουμε και τον συνάδελφο Μάρτιν ε, Κέλναν, ο οποίος είναι ο ε, αρμόδιος από το ECR και έχει τον λόγο. Μάρτιν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα από την αρχή, αλλά έπρεπε να πάω στην ε, διάσκεψη των Προέδρων επιγόντως να πω πρώτα απ' όλα πως η ομάδα μου υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του εισηγητή να διατηρήσουμε τους στόχους του 2020 όπως προτείνει και η Κομισιόν. Οι φυστάμενοι στόχοι, δηλαδή των 147, όπως συμφωνήσαμε πριν από δύο μόλις ε, χρόνια, νομίζω πως είναι ήδη αρκετά ε, φιλόδοξος ε, στόχος Ξέρω λοιπόν ε, ποια είναι η δυσκολία που υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν το ζήτημα ε, που πρέπει να ισορροπήσουμε αφενός ε, της ανάγκης του περιβάλλοντος και από την άλλη βεβαίως και οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν ένα φιλόδοξο στόχο και πρέπει να δούμε βεβαίω και τυχόν περαιτέρω ωφέλη σε συνδυασμό με το κόστος και αντιλαμβάνουμε πως η συμφωνία του 2011 το επέτυχε αυτό. Μάλιστα, μία μελέτη του Βρετανικού Υπουργείου Μεταφορών εκτιμά πως θα εξοικονομηθούν πάνω από 50 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2032. Αν λοιπόν αλλάξουμε τώρα κάτι στη μέση θα υπονομεύσουμε τον σχεδιασμό των βιομηχανιών στη μέση της οικονομικής κρίσης και θα εμποδίσουμε την ανταγωνιστικότητα σε καιρού ε, δυσκολου. Και επίσης, όπως λέει και ο εισηγητή, ε, στο επεξηγηματικό σημείωμα, το περαιτέρω κόστο ε, θα το πληρώσουν ειδικά οι καταναλωτές και πιο συγκεκριμένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγοράζουν τέτοια οχήματα. Όσον αφορά τώρα τα γιοταχή, θα πρότεινα εγώ κάποια σύνεση όσον αφορά την ε, πρόταση αντικατάστασης του κύκλου δοκιμών του παγκόσμιου εναρμονισμένου, καθώς μπορεί έτσι να επηρεαστούν κατά πολύ οι μέθοδοι υπολογισμού στόχων του 2020 και δεν μπορούμε νομίζω και τον κύκλο να τον αλλάξουμε στη μέση της διαδικασίας. Άρα συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να περάσουμε από τον ε, Δεκέμβριο 2014 στην ερήτρα αναθεώρηση ε, του 2018 και να παραμείνει αυτό ως όρος αναφοράς για το στόχο του 2020 αντί να ορίσουμε νέους στόχους βιαστικά. Ανταυτού πρέπει να εστιαστούμε στην, ε, στο σωστό πλαίσιο μετά το 2020 βασιζόμενοι σε πιο καλά δεδομένα. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Κομισιόν προτείνει την παρέκκληση για τους κατασκευαστές ε, μικρών ε, αριθμών, καθώς ε, οι κατασκευαστές που κατασκευάζουν λιγότερα από 500 οχήματα κατ' ουσίαν δεν έχει διαφορά στην μείωση του εξουσίου του άνθρακα, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό των πωλήσεων κάτω από 0,1% και ακόμη λιγότερο αυτού όσον αφορά τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Αντιθέτω, θα επιφέρει σε αυτέ τι μικρέ εταιρείε μεγάλα διοικητικά βάρη. Οπότε η Κομισιόν με αυτή και άλλε προτάσεις για περισσότερη ευελιξία αποδεικνύει πώ αντιλαμβάνεται τις ε, ανάγκε να ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκε των ενδιαφερομένων. Ευχαριστώ, Ζήλ Πανιό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κανονισμός έτσι όπως μας παρουσιάζεται σήμερα είναι κάτι το οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Μέσα σε 20 χρόνια οι εκπομπές αυτού του τύπου των μεταφορών αυξήθηκαν κατά 26%. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τη σωστή πορεία, θα πρέπει να προσανατολίσουμε σε σωστή κατεύθυνση τις εκπομπές αυτών των οχημάτων και να προχωρήσουμε σε μετρήσεις βιομηχανικές και τεχνικές που να επιτρέπουν να υπάρχει καινοτομία και παραγωγή σωστών καθαρών αυτοκινήτων. Και θα συμφωνήσω εδώ με τον συνάδελφο Φλόρεντς στην ανάλυση την οποία έκανε. Θα πρέπει φυσικά στα πλαίσια των προτάσεών μας να μπορέσουμε επίσης όχι μόνο να υποστηρίξουμε, να επιδιώξουμε κάποιους φιλόδοξους στόχους, αλλά να προασπιστούμε και τα συμφέροντα των κατασκευαστών των μικρομεσαίων ε, αυτοκινήτων. Δεν θα πρέπει να υπακούσουμε μόνο σε κριτήρια και επιταγές ε, οικονομικά, αλλά και βιομηχανικά τεχνικά. Οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών έχουν την δυνατότητα ε, να ανταποκριθούν στους στόχους τους οποίους εμείς θέτουμε. Επιτρέψτε μου επίσης να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για το κείμενο. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε το κριτήριο του όγκου του αυτοκινήτου σαν κριτήριο το οποίο δεν συνεισφέρει στην ελάφρυνση του αυτοκινήτου και δεν μειώνει το επίπεδο εκπομπών. Θα κάνω κάποιες προτάσεις μέσω τεχνικών τροπολογιών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το σύνολο τεχνικών προδιαγραφών του 2009 και όχι του 2006, έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή κατανομή ανάμεσα στους κατασκευαστές ε, ε, της προσπάθειας μάλλον ανάμεσα στους κατασκευαστές και θα πρέπει επίσης να υπάρξει και μια χρονική προθεσμία για μετά το 2020 και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος του 2014 να κάνει μια σφαιρική πρόταση σχετικά με την αναθεώρηση του κύκλου ελέγχων έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το σύστημα εκπομπών ευρώ αλλά και ε, το σύστημα ανακοίνωσης και μετάδοσης ε, των ε, αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών. Ευχαριστώ. Γιάννα Ρόσπαχ έχει το λόγο. Όχι. Δεν θέλετε. Κυρία, κυρία Μέρκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να πω κάποια πράγματα. Πρέπει να έχουμε ε, μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως μέχρι και το 2025 και να δούμε τι θα γίνει μέχρι το 2030 και 2050. Και θα βεβαίως θα πρέπει να προσφέρουμε, όπως είπατε, και την ασφάλεια στους κατασκευαστές. Αυτό θα γίνει με το να θέσουμε ένα στόχο μέχρι το 2025. Και για να είμαι ειλικρινής, ε, όπως είπαμε, απέχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά χρόνια και θεωρώ πως τα αυτοκίνητα θα γίνουν ακόμη πιο οικονομικά και κατά την απόψή μου ε, θα πρέπει να έχουμε πραγματικά φιλόδοξη στόξη, η οποία όμως είναι εφικτή. Βλέπουμε πως ε, το σύστημα των super credits δεν θα δουλέψει όπως το θέλουμε. Αντιθέτως, βλέπουμε λοιπόν πως θα επιτευχθεί μια ισορροπία γιατί αυτή τη στιγμή αντισταθμίζονται τα αυτοκίνητα τα οποία καταναλώνουν λίγο. Είτε θα γίνει λοιπόν ένα σύστημα bonus μάλους, είτε κάποιο ίδιο σύστημα πιστώσεων, γιατί έχουμε ένα 50% κακό να πούμε, που θα πρέπει να πληρώνουν το 50% των καλών με κάποιο ε, τρόπο και με ένα σύστημα ETS, ε ETS ε και όπως είπαμε, μια κατεύθυνση η οποία θα είναι προς πιο ακριβά δικαιώματα εκπομπών. Και το μιλάμε για την καινοτομία. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, νομίζω, ειδικά με τα αυτοκίνητα και το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες στο Ρασβούργο όταν μιλούσαμε για τα επίπεδα θορύβου. Και φοβόμαστε πως ε, Εάν δεν έχουμε αρκετά φιλόδοξους ε, στόχους, ε, δεν θα βοηθήσουμε την αυτοκινητομηχανία. Η αυτοκινητομηχανία βοηθιέται με το να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Έτσι δημιουργείται καινοτομία. Αυτό ακριβώς είμαι κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κρίστα Κλάς. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση του κυρίου Κράμερ. Γιατί τι συζήτηση κάναμε και πριν από δύο χρόνια ή τρία. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να βάζουμε καινούριο στόχο και απορώ δηλαδή με αυτά τα οποία, από τα οποία ακούω από τον Καρλ Σλούτερ και την Κορή Λεπάζ, δηλαδή να κάνουμε κάτι για την αυτοκινητοβιομηχανία. Μα ε, ε εντάξει, αυτό θέμε και εμείς. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, το, το είχα πει τότε και θα το πω και σήμερα. Μιλάμε για χειρόνακτες, ε, μιλάμε για εινοποιούς ε, ανθρώπους που πάνε στη δουλειά τους με τα μάξι δηλαδή, όχι βόλτα. Για τα δε όρια ταχύτητας ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους στόχους και να τους τηρούμε γιατί άμα κάθε χρόνο ερχόμαστε και τα αμφισβητούμε, ε, δεν είναι στόχος μετά αυτό. Ποια αξιοπιστία έχουμε. Και η βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι για τις νέες αγορές να έχουμε αυστηρότερες απαιτήσεις. Αλλά ο χρόνος χρήσης μετά πρέπει να ε, είναι μεγάλος για να κάνουν και απόσβεση τα οχήματα, έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ υπήρξα στο παρελθόν σκιώδης εισηγητής για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι είναι κάπως λανθασμένος ο τίτλος αυτής της έκθεσης γιατί πρέπει να μιλάμε περισσότερο για την αποδοτικότητα των, ε, της χρήσης των καυσίμων. Για όλα αυτά όμως θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη αίσθηση ο απλός καταναλωτής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντίφαση εσωτερική στα διάφορα μέτρα και θέλουμε να έχουμε ένα κύκλο δοκιμασίας ο οποίος πράγματι να αντικατοπτρίζει την χρήση που γίνεται από τους καταναλωτές. Ο καθένας έχει μια διαφορετική χρήση των οχημάτων αυτών όταν φτάσουμε όμως σε μια απόκληση 25-30% τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό έχει νόημα σε ένα κύκλο. Για τα super credits επίσης, όπως είπε και ο Καλ θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο και ίσως από τις πολιτικές ομάδες να μπορέσει να προκύψει μια καλύτερη συμβαστική πρόταση για το θέμα αυτό. Γιατί ο στόχος αυτών των πριν των super credits, θα πρέπει να είναι να δώσει κίνητρα, αλλά δεν πρέπει να ανοίξουμε μια κερκόπορτα η οποία θα υπονομεύσει τους στόχους στους οποίους έχουμε θεσπίσει. Και επομένως θα πρέπει να έχουμε και κάποιο ανώτατο όριο για όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει και η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η μικρότερη κατανάλωση σημαίνει και λιγότερα σωματίδια τα οποία πρέπει να εκπέμπονται, λιγότερα οξύδια του αζότου και όλα αυτά επομένως θα πρέπει να μειωθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί και η χρήση καυσίμων, η κατανάλωση καυσίμων. Όλα αυτά σημαίνει ότι θα προκύψει πρόσθετο κόστος, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ των ε, ε, απλών αυτοκινήτων και των ε, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Αν μπορέσουμε όμως να μειώσουμε το κόστος χρήσης, δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση, αυτό πρέπει να είναι το κύριο επιχείρημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και έχει νόημα να προχωρήσουμε σε καινοτομίες οι οποίες θα μειώσουν αυτή την κατανάλωση. Επίση, στη συζήτηση πριν από δύο χρόνια, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, είχαμε θέσει και το θέμα των περιοριστών ταχύτητων, των κοπτών όπως λέμε. Ο πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση της κατανάλωση είναι το να μην κινείται κανείς με υψηλή ταχύτητα. Επομένως για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Τότε είχαν ψηφίσει υπέρ οι συνάδελφοι για την Επιτροπή, στην Επιτροπή Μεταφορών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος βέβαια είχε απορρίψει αυτό το μέτρο. Θα πρέπει όμως να δώσουμε τη δυνατότητα και στα super credits για τα κάτι μελη που το επιθυμούν να δώσουν και φορολογικές απαλλαγές για οχήματα τα οποία θα είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον. Δηλαδή για τα οχήματα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση, θα πρέπει τότε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάποιο μπόνους σε επίπεδο φορολογικής μεταχείρισης για τα οχήματα αυτά και σε ό,τι αφορά τους πιο ε, μακρόπνοους στόχους που μας ενδιαφέρουν. Εδώ έχει δίκιο και ο κύριος Κράμερ και η συνάδελφοι ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να έχει κάποια σταθερότητα σε σχέση με τις συνθήκες για να κάνει σωστή σχεδίαση. Θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε κύκλους σχεδιασμού και παραγωγής της τάξεως των 7 ετών, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ορίζοντα που να μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίε χωρίς υπερβολικές δυσκολίες. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο θα πρέπει να είναι ο μακρόπνος στόχος που θα γίνει αποδεκτός. Σίγουρα σε τελική ανάλυση το να υπάρξει η μείωση της κατανάλωσης. Αυτό βοηθάει το μαραγκό, βοηθάει τον ε, ε, αμπελουργό, βοηθάει όλους αυτούς να έχουν μικρότερο κόστος στις επιχειρήσεις τους αν τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν θα είναι πιο οικονομικά και μπορούν με τον τρόπο αυτό να επιτύχουν εξοικονομήσεις. Για μένα από τα πιο σημαντικότερα στοιχεία είναι ακριβώς η βελτίωση του κύκλου δοκιμασιών. Αν λοιπόν έχουμε οχήματα τα οποία άλλα αποτελέσματα βγάζουν στον κύκλο δοκιμασίας και 20-30% περισσότερο σε πραγματική χρήση, αυτό δεν έχει κανένα όνομα. Θα πρέπει να μην υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση και το πολύ πολύ μπορούμε να δεχτούμε ίσως μια απόκληση της τάξης 10% αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα απεριόριστο επίπεδο ε, απόκληση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόν, ο οποίο είναι ο επικεφαλή μονάδα, ο αρμόδιο για τα θέματα αυτά τη ε, αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω και τον κύριο Κράμερ για την έκθεση αυτή που περιέχει μια πλειάδα νέων ιδεών. Να ξεκινήσω με μερικά πραγματικά στοιχεία. Ο στόχος του 2010 ήταν 180 Μάλλον το στοιχείο το πραγματικό ήταν 181 γραμμάρια το 2010 και θέσει πίσω το Κοινοβούλιο ένα στόχο για 175 γραμμάρια το 2017 και όπως ξέρει και ο κύριος ε, Φλόρενς μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στο στόχο του 147, γραμμα, το 147 γραμμαρίων για το 2020 και γι' αυτό εκπλήσωμε για τις τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται στην έκθεση αυτή και θέλουν ήδη να τροποποιήσουν αυτούς τους στόχους. Με τα super credits έχουμε ήδη αλλάξει τα επίπεδα συμμόρφωσης και το ανώτατο όριο για τα οχήματα επί τη βάση του στόχου 175 γραμμαρίων για το 2017, όταν σήμερα είμαστε μονάχα στα 100, είμαστε στα 181. Ε, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί ο στόχος του 147, του 175 καταρχήν, υπονομεύεται. Ο στόχος του 147 τα γραμμαρίων, αυτός πιστεύω ότι είναι εφικτός, πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε με λογικό κόστος για την βιομηχανία. Και πάλι αυτός ο στόχος, πέραν αυτών που ελέγχθηκαν, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί με νέους πολλαπλασιαστές, με νέα κατόφλια για τα Super ή με το να αυξήσουμε την οροφή του αριθμού οχημάτων που καλύπτονται. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια διαδικασία συσσόρευσης που θα επιτρέψει τα πρίμα αυτά να συσσωρεύουν το 2019. 2020 και να εφαρμόσουμε στη συνέχεια. Κάναμε κάποιους υπολογισμούς για το τι μπορεί να γίνει. Αν 2% των οχημάτων των ελαφρών επαγγελματικών καλύπτονται από τα ε, super credits, τότε ο στόχος θα ανέβει στο 152. και δεν θα έχουμε κάτι χαμηλότερο από το 147 το 2025. Η αλλαγή λοιπόν αυτών των στόχων θα οδηγήσει στα... σε μια μείωση των αποτελεσμάτων μετρίασης της κλιματικής αλλαγής με να αυξήσει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Πολλοί αναφέρθηκαν επίσης και στον κύκλο δοκιμασιών να ξεκινήσω τονίζοντας κάτι το οποίο είναι σαφές στη δική μας πρόταση. Αν ο κύκλος δοκιμασιών αλλάξει και χρησιμοποιήσει τα πρότυπα WLTP, εμείς έχουμε αναλάβει να κάνουμε την απαραίτητη προσαρμογή και να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι πιο ε, αυστηρός αυτός ο κύκλος για τους κατασκευαστές. Ό,τι και να γίνει λοιπόν, ο κύκλος θα παραμείνει ο ίδιος. Δεν θα αλλάξει τίποτα η μετάβαση από το NEDC στο WLTP. Δεν θέλουμε να οδηγήσουμε σε πρόσθετο άχθος για τους κατασκευαστές μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Είναι σημαντικό όμως να ενσωματώσουμε το νέο κύκλο WLTP. Η διαδικασία του NDC e θα φτάσει μέχρι το 2013 από το 2014 θα γίνει η αντικατάσταση και θα εφαρμόζεται ο κύκλος WLTP. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό δίνουμε καλύτερη πληροφόρηση στους αγοραστές των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι καταναλώνουν τα οχήματά τους οι αγοραστές και αυτό θα επιτρέψει να υπάρχει καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων και αν υπάρξει κόστος για να επιτευχθεί ο στόχος του 147 θα μπορούν να δουν οι ιδιοκτήτες των ελαφρών απογευματικών οχημάτων από τη χρήση των γνωρίζοντας σε ποιο κομμάτι της χρήσης θα μπορεί να προκύψει η εξοικονόμηση. Νομίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν όλους στη διαδικασία αυτή και αντί να έχουμε πρόσθετο κόστος θα έχουμε πραγματικά εξοικονόμηση για τους αγοραστές των νέων αυτών οχημάτων. Και έρχομαι τώρα στους μακροχρόνιους στόχους και για το πότε θα πρέπει να διατυπωθούν αυτοί οι στόχοι. Εμείς προτείνουμε το 2014 γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται το χρόνο σχεδίασης και το χρόνο προσαρμογής. Χρειάζονται μια βεβαιότητα. Το να καθυστερήσουμε την θέσπιση των στόχων για τέσσερα χρόνια θα κάνει τα πράγματα μόνο χειρότερα. Θέλουμε να είναι ανταγωνιστική η αυτοκινητοβιομηχανία μας. Το ταχύτερο που θα φέρουμε αυτούς τους στόχους είναι μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα που θα έχουν οι βιομηχανίες για να κάνουν την απαραίτητη προσαρμογή και να μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους που επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Χόλγκερ Κράμερ, ο συζήτης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τα επιχειρήματα. Υπάρχουν διάφορες πτυχές. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα σημαντικότερα που θα για τον κύκλο δοκιμών Βεβαίω, αγαπητέ Καλ Χάιντς, Φίλιπ Όουεν και λοιποί, ο κύκλος ε, δοκιμών δεν είναι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι πως ο κύκλος αυτός δεν είναι αντικείμενο του κανονισμού μας. Είναι άλλο το θέμα της συζήτηση σήμερα. Ανεξαρτήτως του πώς έχει λοιπόν αυτός ο κύκλος, είναι ε, ένας τρόπος να είναι συγκρίσιμα τα οχήματα και να ορίσουμε στόχους του διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε εγώ δεν έχω στόχο εδώ πέρα να αλλάξω τον κύκλο δοκιμών. Αλλά τι λέω, όταν θα έχουμε νέο κύκλο, τότε θα πρέπει να ορίσουμε νέο μακροπρόθεσμο στόχο. Εάν δεν έχουμε και υπάρχει μια κάποια πιθανότητα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι να μην καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία, πρέπει να είναι ξεκάθαρο και για λόγους προγραμματισμού ότι θα συνεχίσουμε με τον παλιό. Τώρα, αν θα έχουμε έναν δικό μας ευρωπαϊκό, και αυτό αξίζει να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι αντικείμενο αυτού του κανονισμού. Θεωρώ πως πρέπει να πω αυτό το οποίο είπαμε και στην Επιτροπή ε, Βιομηχανία και που ισχύει και για τα ΙΟΤΑΧΗ, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ε, κατασκευαστών που ε, έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό, πολύ χαμηλό, με συγχωρείτε, πολύ του άνθρακα και αγοραστικής επιτυχίας. Ισχύει μάλιστα το αντίστροφο. Αυτοί που φτιάχνουν μικρότερα αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπέ δεν σημαίνει πως αυτομάτως έχουν τις καλύτερες πωλήσει. Είναι παρεξήγηση αυτή τη συζήτηση και θέλω να σας το πω. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι υποστηρίζουν έτσι τη βιομηχανία. Εγώ δεν θέλω να πω στη βιομηχανία πώς θα φτιάξει τα αυτοκίνητά της. Αυτό το ξέρει, όποιος το ξέρει καλύτερα από τη βιομηχανία μπορεί να ανοίξει δική του αυτοκίνητο βιομηχανία πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο νομικό πλαίσιο βεβαίω. Θεωρώ, για να το ξαναπώ, πως το 2014 είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε και να πούμε το τι θα γίνει μετά το 2020. Γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, συμβαίνουν πάρα πολλά είδη, τόποι και online. Εμφανίζονται νέες τεχνολογίες στους κινητήρες, δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα επικρατήσει, μειώνονται οι τιμές της, ε, του φυσικού αερίου, μπορεί να έχουμε φυσικό αέριο. Γιατί θα είναι πολύ φτηνότερο. Ε, απλά δεν το ξέρουμε σήμερα. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε λίγο χρόνο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στις αγορές. Μια συμβιβαστική πρόταση. Να μην είναι το 2018, αλλά το 2014 είναι πολύ νωρίς θεωρώ. Οι πιστώσεις αυτές, ε, τα super credits. Ναι, δεν είναι... Να τα αλλάξουμε το όνομα, δεν είναι πιστός που πληρώνει ο φορολογούμενος, μπορούμε να το πούμε ε, κίνητρο καινοτομία. Βλέπω πως ε, θέλουν κάποιοι να παραμείνει στον τομέα των ελαφρών οχημάτων. Τώρα, αν θα υπάρξει κάποιο όριο ή όχι, θα το αφήσουμε. Οι κόφτες επίσης δεν κολλάνε εδώ σε αυτόν τον οργανισμό. Και δεν είναι και ο αποτελεσματικότερο ε, τρόπο μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, κύριε Πρόεδρε. Άμα είναι έτσι, δηλαδή ο αποτελεσματικότερο τρόπο είναι να μην βάλουμε καν μπροστά το αυτοκίνητο. Δεν είναι η δική μα η δουλειά. Να πούμε σε ανθρώπου που 100% χρησιμοποιούν το όχημα για τη δουλειά του, έτσι. Όχι για... για άλλο σκοπό. Να, να τους εκνευρίζουμε. Γιατί τελικά έτσι δημιουργείται και πρόβλημα οδική ασφάλεια. Δεν πρέπει αυτό να το πούμε, να το ορίσουμε νομοθετικά. Υπάρχουν εξάλλου οι εταιρείε που έχουν μεγάλους στόλου. το, κάνουν μόνοι τους αυτό, βάζουν ένα κόφτη ε, και γίνεται θελοντικά, δεν ανάγκη να το πει ο νομοθέτης. Οι δε μικροί κατασκευαστές ε, δεν πρέπει να είναι νομίζω το βασικό αντικείμενο της συζήτησή μας. Δεν θα μειώσουν. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε συνολικά με το μέσο όρο του στόλου. Αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται, εξαιρούνται δικαίω. Είναι πολύ μικρά τα νούμερα. Χαίρομαι λοιπόν για τη συζήτηση. Ε, για τον δε εκπρόσωπο της Κομισιόν ε, θα σας δείξω τις επόμενες μέρες μια μελέτη που καταλήγει σε άλλο ε, ε, συμπέρασμα από εσά. Δηλαδή λέει πως οικονομικά ρεαλιστικός στόχος πρέπει να είναι μεταξύ 207 και 130 τόσων γραμμαρίων. Δεν σημαίνει το υιοθετώ, απλά δείχνει πως δεν υπάρχει ε, αυτοματισμός, εάν θέλετε, ότι φιλόδοξη νομοθεσία ε, όσον αφορά το εξίου του άνθρακα ε, ωφελεί τον καταναλωτή. Υπάρχει πάντα κόστος. Ε, κόστος ανάπτυξης οχήματος, ε, τελική τιμή, κάποιος το πληρώνει αυτό στο τέλος. Και η κυρία Γκροστέτ είπε σωστά πως αν τους δημιουργήσουμε προβλήματα θα αγοράσουν μεταχειρισμένα φορτηγά και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση. Νομίζω λοιπόν πως έχουμε κατάληξει έναν ικανοποιητικό συμβασμό. Φιλόδοξοι λοιπόν νομίζω ότι είμαστε, αλλά και ρεαλιστές σας παρακαλώ για να μην ε, πλήξουμε την ε, αυτοκινητομηχανία, ειδικά καθώς ο Νότος Ευρώπης δεν βρίσκεται και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 27 Φεβρουαρίου 12 η ώρα. στις 25 Απριλίου θα τη συζητήσουμε στην Επιτροπή, 6 Μαΐου ψηφοφορία και στην Ολομέλεια θα πάει ενδεικτικά ε, στην Ολομέλεια του Ιουλίου 2013. Άρα τελειώσαμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο επόμενο. Περνάμε στην πρόταση λοιπόν ε, Stop the Clock τη λεγόμενη, την προσωρινή παρέκκληση. Συγητής είναι ο Πέτερ Λίζε. Του δίνω το λόγο να μας κάνει μια εισαγωγή. Yeah, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα συζητήσουμε μονάχα για τις τροπολογίες και εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουν ε, υποβληθεί πολλές τροπολογίες οι οποίες ακολουθούν την οδηγόγραμμη του εισηγητή και βελτιώνουν το έγγραφό μου. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών με εισηγητή το Μάτιου Γκρός που έχει κάνει σημαντική και επικοδομητική συμβολή για τα θέματα αυτά και ελπίζω θα μπορέσουμε σήμερα να προετοιμάσουμε μια συμφωνία με την Επιτροπή Μεταφορών ενώπιον της ε, ψηφοφορίας που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Για αυτούς που δεν ήταν παρόντες την τελευταία φορά, να κάνω μια γενική επισκόπηση για αυτά που έχουν λάβει η χώρα. Η Κομισιόν έχει προτείνει πριν από να διατηρήσουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2014 το καθεστώς για τις ε, αεροπορικές πτήσεις. Δεν θα υπάρχει λοιπόν καμία κύρωση σε όχι σε σχέση με τις ε, πτήσεις οι οποίες ξεπερνούν τα όρια αυτά. Αυτές οι εξαιρέσεις λοιπόν εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις ε, διυπηρωτικές πτήσεις, όχι μοναχά τις Ευρωπαϊκού, από των ευρωπαϊκών εταιριών, όλες αυτές οι οποίες έρχονται στην Ευρώπη ή πηγαίνουν στην Ευρώπη ξεκινώντας από μια τρίτη χώρα ή φεύγουν από την Ευρώπη ή πηγαίνουν δηλαδή στην Ευρώπη. Για τις ενδοευρωπαϊκές ε, πτήσεις αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί μαζί σας, αλλά νομίζω ότι ο στόχος μας τελικά είναι να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν θα κάνει καμία διάκριση μεταξύ Ευρώπης, ε, Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας κτλ. Είναι πολύ καλό να περιορίσουμε κάθε μορφή εξαιρέσεων και χρονικά και σε επίπεδο ουσίας. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια διεθνή συμφωνία. Θέλουμε όμως να διατηρήσουμε το σύστημα αυτοεμπορίας εκπομπών και όλα αυτά να μεταβληθούν σε μια παγκόσμια συμφωνία. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν και νομίζω ότι είναι καλό σημείο εκκίνησης. Υπάρχει βέβαια και το ερώτημα γιατί υπάρχει αντίσταση από τόσα πολλά τρίτα κράτη. Εδώ θέλω να κάνω σαφές ότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν πραγματικά επιχειρήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί. Είναι ουσιαστικά ένα πολιτικό παιχνίδι γιατί είναι πραγματικά πολύ περιορισμένη η επιβάρυνση η οποία αφορά τις διπηρεωτικές πτήσεις. Πρόκειται για κάθε επιβάτη για 2 ευρώ και αυτό είναι πολύ λιγότερο από αυτό που πληρώνει κανείς στο αεροδρόμιο για ένα καφέ και επίσης το θέμα ότι παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των ε, τρίτων χωρών για την εμπορία εκπομπών. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει ως επιχείρημα με μεγάλη γαλήνη, γιατί ήταν σαφές από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι έχουμε την δυνατότητα να, βάλουμε, να επιβάλλουμε τέλη για αεροπλάνα τα οποία ε, προσγειώνονται ή απογειώνονται από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ε, ούτω ή άλλως δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτά τα, οποία, τα τέλη τα οποία επιβάλλονται στα γερμανικά και τα αγγλικά αεροδρόμια. Όταν πετάει τώρα μία ε, μια αεροπορική εταιρεία από την ε, Γερμανία ή στην Πολωνία ή από την, είναι, είναι φτηνότερα από ότι για την, ε, πετάει μια εταιρεία από την Αγγλία στον Καναδά ή από τη Γερμανία στον Χογκό κτλ. Επομένως αυτό το επιχείρημα των τρίτων κρατών δεν στέκεται. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταλάβουμε ότι είναι αποφασιστική η απο τη γερμανια στον χογκο κτλ επομενως αυτο το επιχειρημα των τριτων κρατων δεν στέχεται. ειναι απαραιτητο λοιπον να καταλαβουμε οτι ειναι αποφασιστικη η αντιληψη που υπάρχει. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν του ενδιαφέρει να υπάρξει μια διεθνή ρύθμιση για τα θέματα αυτά και χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα για να το εμποδίσουν. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω τι προτάσει τη Κομισιόν στην ουσία τους και γι' αυτό οι τροπολογίες οι οποίες αποκλίνουν από την πρόταση της Κομισιόν σε ουσιαστικό επίπεδο για μένα δεν πρέπει να γίνονται δεκτές. Οι τροπολογίες 8 της Βίλτς και Σατου δεν είναι παρούσες, αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι οι σοβαρές ενώσεις για το περιβάλλον, όπως και η σοβαρή βιομηχανική ε, βιομηχανικό χώρο δεν δέχονται αυτές τις ε, προτάσεις της κυρίας Χάση και Βίλς. Και δεν ξέρω αν και οι ίδιες οι συγγήτριες θέλουν να γίνουν δεκτές τέτοιου είδους ε, τροπολογίες όπως αυτές έχουν προτείνει. Γι' αυτό θα ήθελα να τις παρακινήσω να αποσύρουν αυτή την τροπολογία. Γιατί τροπολογίες 11 και 20 έχουν αποσυρθεί. Εδώ πρόκειται για μια καθυστέρηση κατά ένα χρόνο για την ημερομηνία εφαρμογής, δύο χρόνια αντί για ένα. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θέλουν να εξασφαλίσουν με αυτές τις τροπολογίες. Ή θα γίνει η εφαρμογή με τον τρόπο αυτό που προτείνεται από την ΙΚΑΟ ή δεν θα καταλήξουμε σε καμία συμφωνία. Σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια λύση που θα οδηγήσει στο να ισχύει το σύστημα εκπομπών μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην καλύπτει τις διυπηρωτικές πτήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο διεθνής, διεθνούς και αν το κάνουμε αυτό μόνο μετά από δύο χρόνια δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τον ορίζοντα 2022 και θα έχουμε και ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Η, η, το κόστος για, την, για τις εκπομπές αυτές θα είναι πολύ χαμηλό. Παραγματικά η Φραγκφούρτη, Αμβούργο 13 σεντ μονάχα. Αλλά ε, δεν θα υπάρξει καμιά λύση για τις διεθνείς πτήσεις, γι' αυτό απορρίπτω τις τροπολογίες 11 και 20. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες οι οποίες εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σαφήνεια και θέλω να τις υποστηρίξω. Καταρχήν μια τροπολογία του Προέδρου και της κυρίας Μπράντι, και Μπράντι. Όλες αυτές θα μπορούν να περιληφθούν σε μια συμβαστική λύση. Υπάρχουν επίσης τρεις τροπολογίες που θεωρώ ότι είναι σημαντικές γιατί καλύπτουν και νέες πτυχές της συζήτησης που έχουν ανακύψει και νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Πρόκειται για το λεγόμενο earmarking, τον προσδιορισμό και είναι αυτές οι οποίες προέρχονται από την Επιτροπή Μεταφορών με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα τα οποία θα εισπραχθούν από αυτά τα μέτρα θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο λύση τελή για να προωθήσουμε την τεχνολογία και την ε, καινοτομία με την έρευνα στις αεροπορικές βιομηχανίες. Υπάρχει επίσης τροπολογία Χασί και Βίλς και η δοπική μου τροπολογία 30 που αφορούν την ε, έγκριση από τρίτα κράτη. Αν συμφωνήσουν οι Αμερικανοί παραγωγός μπορούμε να κάνουμε με ένα τμήμα αυτών των ποσών που θα εισπραχτούν κοινά προγράμματα έρευνας. Και επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε τα χρήματα αυτά για την υποστήριξη της κλιματικής ε, πολιτικής μέσω ενός Ταμείου Παραγματος Χάρη του ΟΗΕ. Αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει και σε μια πιο εύκολη έγκριση των ε, τρίτων χωρών, των αναπτυσσόμενων χωρών. Σας πεθυμίζω ότι έχουμε να κάνουμε και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά που, έχουν, που έχει μέχρι στιγμής απορρίψει αυτές τις κατευθύνσεις, θα πρέπει εμείς με τις θέσεις μας να κάνουμε σαφές σε παγκόσμιο επίπεδο ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε προς το ευρύτερο συμφέρον αυτά τα ποσά και αυτό θα διευκολύνει και την έγκριση αυτών των ε, θέσεων. Καταλήγω λοιπόν στα εξή συμπεράσματα ότι η γραμμή που θέλω εγώ να υποστηρίξω είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε μια λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να αποφευθούν οποιασδήποτε ρυθμίσεις οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι εμείς θέλουμε να ε, θέσουμε στις ελληνικές καλένδες το σύστημα αυτό για την εμπορία εκπομπών και δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα προβλήματα τη εμπορία εκπομπών. πήρα ένα email που έλεγε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το σύστημα του ETS. Πρόκειται λοιπόν όχι μόνο για θέμα τεχνικών ρυθμίσεων, αλλά για το θέμα του αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντησή μου είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το σύστημα αυτό. Αντίθετα, θα πρέπει να ενισχυθεί και πάλι το σύστημα αυτό και κυρίω να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. yes, we can, λέει ο σας ευχαριστώ Πέτερ Λίζε. Αύριο θα, συζητήσουμε, θα αποφασίσουμε για το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε όλοι να εξασφαλίσουμε μια επιτυχία στις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του ΙΚΑΟ και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα μόνο αν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσουμε να είμαστε ενωμένοι. Εδώ και 12 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και το πρόβλημα υπήρξε μονάχα, το πρόβλημα έφτασε στην επιφάνεια μόνο όταν οι Αμερικοί, οι Ηνωμένε Πολιτείες θέλησαν να έχουν το δικό τους σύστημα. Όπως είπε λοιπόν ο εισηγητής, δεν είναι ο στόχος να πάρουμε κάποια χρήματα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να τα χρησιμοποιήσουμε για καλύτερη έρευνα στον τομέα αυτό. Μόνο αυτή η λογική υπάρχει. Γιατί είδαμε πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν θέσει κάτι τέτοια τέλη για πτήσεις οι οποίες είναι πολύ ε, μικρές, πολύ σύντομες, πληρώνουμε 10 φορές παραπτήσεις που είναι πολύ πιο μακρές, που έχουν 10 φορές μεγαλύτερο, μεγαλύτερη απόσταση. Έχουμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα, πράγματι την ευκαιρία αυτή, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μία διεθνή συμφωνία και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την κατεύθυνση, όπως έχει προτείνει και η Κομισιόν, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την ε, υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και να μπορέσουμε να έχουμε μία αποφασιστική τομή στα πλαίσια του ΙΚΑΟ. Και εγώ μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω τη γραμμή του εισηγητή στα θέματα αυτά. Όλα εξαρτώνται από την αυριανή ψηφοφορία βέβαια όπως είπαμε. Αν μπορούμε να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό για την ε, για την τιμή του διοξίδιου του άνθρακος ή αν αντίθετα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή στην ψηφοφορία αυτή για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να διατηρηθεί το σύστημα αυτό για την τιμή του διοξιδίου του άνθρακος. Μπορούμε ούτως ή άλλως να είμαστε υπερήφανοι για όλα αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει για το σύστημα αυτό για τις ε, αεροπορικές πτήσεις και πρέπει να αποφασίσουμε να υπάρχει κάποιο σύστημα ούτω ή άλλω, είτε ένα σύστημα φορολογικού χαρακτήρα, είτε ένα σύστημα εμπορία. Εγώ πιστεύω ότι το ETS είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει καλύτερα και σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό απαιτεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ μα. Έρχομαι τώρα με του ε, επόμενου ομιλητέ, ο Chris Davis. Και έχει το λόγο. Δεν ζήτησα το λόγο. Θέλω να μιλήσω βέβαια. Γι' αυτό ίσως ε, να πάρω το λόγο λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. Καλώς. Μάρτιν Κάλαναν, λοιπόν. Θέλετε τον λόγο. Βεβαίως. Έμα ε, έτσι είναι όταν ο ένας από τον κυβερνητικό συνασπισμό δίνει το λόγο στον άλλον. Είναι ωραία. Θα είμαι σύντομο όπω ακούστηκε και πριν. Η αναβολή για ένα έτος σχετικά με την απόκληση για την εξαίρεση για τις πτήσεις ε, από τις Γενικές Συμφωνίες τις τομεακές θα πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση του ταχύτερο δυνατόν με ελάχιστες τροπολογίες. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αιρεσιμότητα από ό,τι στην προηγούμενη πρόταση και δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την τύχη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογραμμίζω εδώ τις τροπολογίες που θέλουν να ξανανοίξει η συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν σε σχέση με την προσημείωση των εσόδων από τους διαγωνισμούς τους πληστηριασμούς μάλλον των ποσοστώσεων και νομίζω ότι έτσι και αλλιώς τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να δεχθούν το αίτημα αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τις τροπολογίες που προκαταλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις του ΙΚΑΟ και δεν νομίζω ότι χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρξουν επιπλέον προϋποθέσεις ειδικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τους στόχους και σε σχέση με ε, τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να το πετύχουμε. Θα πρέπει επίσης ε, να αποκλείσουμε κάποιες γραφειοκρατικές διατυπώσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα ε, στους διαπραγματευτές οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους το ταχύτερο δυνατόν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία ικανοποιητική για όλους τους εμπλεκομένους. Σλούτα έχει ζητήσει το λόγο. Εκπροσωπεί την πολιτική του ομάδα. Θα ήθελα να υπάρξει τέλος αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους μέσα στους οποίους κινούνται τα αεροσκάφη πλέον σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς προτείναμε να απορριφθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Συμφωνούμε όμως με την τροπολογία 23, έχουμε καταθέσει μια παρόμοια και εμείς την 24, όπου ζητάμε εμείς να δοθούν τα έσοδα σε συγκεκριμένους χρήσιμους στόχους, με τους οποίους θα συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουν τα ρολόγια περιμένοντας, θα πρέπει να πιέσουμε για μια σφαιρική συμφωνία προχωρώντας με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και για δράση σε τρίτες χώρες και για την έρευνα και την ανάπτυξη υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν μειωμένες αντιστάσεις και να πετύχουμε την επιθυμητή παγκόσμια συμφωνία. Ήδη ε, υπάρχει ελεύθερη κατανομή κατά 85%. Υπάρχουν πληστηριασμοί μόνο για το 15%. Μιλάμε για το ελάχιστο ε, το οποίο θα πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτικό. Και δεν είναι σωστό νομοθετικά να πούμε ότι θέλουμε εμείς ένα μέσο που να βασίζεται στην αγορά και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του μέσου αυτού να πούμε «Α, όχι, μετανιώσαμε, πρέπει να σταματήσει». Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη της αγοράς. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία για να αναγνωρίσουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενδιαφέρουσα. Το να σταματήσουν οι μετρητές, τα ρολόγια αν θέλετε, περιμένοντας ε, μια θετική απόφαση από πλευρά του ΙΚΑΟ, η οποία ελπίζω να λυθεί το ταχύτερο δυνατόν. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι η οδηγία θα ε, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2012 και ήδη έχει υπάρξει μια πρόταση τροποποίησης από τις 12 Νοεμβρίου. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κάποιες ε, θα έλεγα φάσεις αβεβαιότητας μέσα από τις οποίες ε, κινούνται, στις οποίες κινούνται οι βιομηχανικοί κύκλοι. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς και ποιες είναι οι αναδρομικές επιπτώσεις ε, για τους αερομεταφορείς και για τις επιχειρήσεις γενικά οι οποίες έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Ορισμένοι αερομεταφορείς έχουν ξεκινήσει να αγοράζουν ένα τμήμα των πιστώσεων για τις ε, πτήσεις τις οποίες έχουν εκτελέσει πριν από τις 12 ε, Νοεμβρίου. Ακριβώς ήταν καλοί μαθητές ε, και προκατέλαβαν κατά κάποιο τρόπο το 2013. Έτσι λοιπόν τους δημιουργούμε ένα πρόβλημα γιατί λειτουργεί το σύστημα εις βάρος τους προσπαθώντας να τους πιέσουμε να λειτουργήσουν με τα κριτήρια του 13 ακόμα και το 12. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι στάθηκαν καλοί μαθητές και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη νομική βεβαιότητα των ρυθμίσεών μας, μην επιβαρίζοντας εκ των υστέρων κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται για την πιστοποίηση όλων αυτών των μέτρων. Γι' αυτό προτείνω λοιπόν και μία τροπολογία η οποία θα επιτρέψει την εφαρμογή της οδηγίας ως έχει και ως ήταν γνωστή από τους αερομεταφορείς χωρίς να υπάρξουν ε, μειονεκτικές επιπτώσεις για αυτούς που έχουν ήδη προχωρήσει στην λήψη μέτρων από το 12. Είναι σκανδαλώδες το να ρίξουμε και να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι πήραν τα μέτρα που έπρεπε ήδη από το 12 και εις βάρος τους να λειτουργήσει το σύστημα και υπέρ αυτών που δεν έκαναν τίποτα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να καταλήξει σε ένα θετικό θα έλεγα αποτέλεσμα και να βοηθήσει στη Σφαιρική Συμφωνία στο ΙΚΑΟ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω τώρα να επαναλάβω τη συζήτηση. Εγώ θα ασχοληθώ μόνο με τις τροπολογίες. Το Stop the Clock δεν είναι λανθασμένος τίτλος. Ε, δεν σταματάμε το ρολόι, αλλά πάμε προς τα πίσω. Και είχαμε τεράστια αντίσταση από πάρα πολλές ε, χώρες που δεν αποδέχτηκαν πολύ απλά. Το, θα τους επιβάλλουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό έγινε άρα γιατί δεν υπήρχε λύση. Και αυτό το κάνουμε με μισή καρδιά. Γιατί οι πτήσεις ε, προς τρίτες χώρες δεν ε, υπάγονται στο δικό μα το σύστημα, το ETS. Τώρα ε, ακριβό φτηνό είναι διάφορο. Να σας το πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι πήγα από τον Ντίσσελτοφ στην Μαγιόρκα. Είναι στο ETS μια πτήση από το Düsseldorf στην Αίγυπτο δεν είναι στο ETS. Και ε, αντιλαμβάνεστε βεβαίω πόσο ευαίσθητοι είναι οι τουρίστες και τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορία. Τι μπορεί κάλλιστα να σημάνει αυτό α, κέρδος για την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένη περίπτωση και τα αιγυπτιακά θέρετρα Έτσι, χωρίς όφελος για το κλίμα. Οπότε, εγώ ε, έχω ε, υπογράψει την τροπολογία που λέει εάν είναι ε, να έχουμε το ETS ε τότε συνολικά, όχι για λόγους φιλοδοξίες, αλλά για το Yes το οποίο είπες και το οποίο δεν το έχουμε. Δηλαδή μπορεί στον ΙΚΑΟ το φθινόπωρο να μην γίνει τίποτα. Τι θα κάνουμε τότε. Πάλι θα είμαστε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε πολιτικές συγκρούσεις, ε, ε, επιστολές υπουργών εξωτερικών και άλλα τέτοια παρόμοια και θα έχουμε πάλι το αδιέξοδο που είχαμε και πέρσι. Δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό. Πρέπει, ακόμα και αν καταλήξουμε σε έναν αποτέλεσμα το φθινόπωρο, να έχουμε την ε, δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια νομοθετική εφαρμογή των όσων αποφασιστούν στον ΙΚΑΟ. Μπορεί κάλλιστα να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μπορεί και να μην προκύψει τίποτα, όπως είπα και να έχουμε μια ευρωπαϊκή νησίδα που κάτι μόνο θα κοστίζει και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί, το είπε και ο Πέτερ Λίζε έτσι γρήγορα, τότε εάν κάνουμε κάτι για όλους. Έτσι. Ε, ή και αν το αναβάλουμε επίσης, να το αναβάλουμε επίσης για όλους. Και είναι ένα ζήτημα, όπως είπα, διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να βγουν εκτός αυτή τη στιγμή τα, οι τρίτες χώρες. Οι χώρες όμως εζές που δεν ε, υπερψήφισαν ε, το ETS, ε, το να τους το επιβάλλουμε είναι μια πρόκληση άκυρη και άχρηστη. Έτσι. Και παριστάνει η Ευρώπη τη δυνατή εδώ πέρα απέναντι σε αυτές τις χώρες. Και πραγματικά Ορμάμε σαν ε, τάβρος ε, ενιαλοπολείο στο διπλωματικό επίπεδο. Η Ελβετία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να του υπαγορεύουμε τι θα κάνουν. Έτσι. Υπάρχει το διεθνέ δίκαιο. Τουλάχιστον οι χώρε ΕΖΕΣ που δεν συμφώνησαν δεν μπορούμε να τι εξαναγκάσουμε. Ευχαριστώ, Βέσλοντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Θα είμαι σύντομη. Για μένα μου φάνηκε κάπως παράξενη αυτή η πρόταση από την Κομισιόν όταν διατυπώθηκε στην αρχή. Εγώ άκουσα ένα επιχείρημα για την υποστήριξη της Κομισιόν, δηλαδή το ότι δεν μπορούμε να χρονοτριβήσουμε πάρα πολύ σε επίπεδο εφαρμογής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση και, καταλήξουμε σε μια, και να καταλήξουμε σε μια κατάσταση μόνο ασαφών υποσχέσεων. Όπως είπε και ο Πέτερ Λίζε, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και επομένως αυτό είναι μια καλή στρατηγική. Θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, αλλά αυτό απαιτεί μια σαφή καθοριστική, καταληκτική ημερομηνία που δεν πρέπει να απέχει πολύ στο μέλλον και να έχουμε και συγκεκριμένα κριτήρια. Και αν δεν υπάρξει καμία πρόοδος θα πρέπει να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα ETS. Και φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βάρος που επιβάλλουμε σε αεροπορικές εταιρείε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πετάμε τόσο πολύ. Όλο και περισσότερο πετάνε οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στο διηνεκές. Αν μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να περιμένουμε για να επιτευχθεί, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα. Αν δεν υπάρξει λοιπόν κάποια λύση, θα, καλύπτει θα πρέπει να καλύψουμε μόνο τις ευρωπαϊκές πτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κριστέβης και πάλι. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και απλός. Συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει κάποιος χώρος για διαπραγματεύσεις Θέλω όμως ε, να μην υπάρξει προσημείωση των συγκεκριμένων εσόδων από τους πληστηριασμούς και να θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή, εν πάση περιπτώσει. Στην περίπτωση σαν παράδειγμα των κινητών κλιματιστικών μονάδων λέει ότι εμείς διακόπτουμε την ισχύ της νομοθεσίας για δύο έτη. Μπορεί να το κάνει αυτό θεωρητικά βέβαια και μπορεί να το τεκμηριώσει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν επιχειρήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά θα πρέπει να ομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει ανάγκη για κάπως μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χώρο. Και δεύτερον, ε, με τη συζήτηση αυτή δεν καταλαβαίνει κανείς που ακριβώς βρισκόμαστε. Απλά λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις και ακόμα και αν υπάρχει ένας χρονισμός προαποφασισμένος, οι συζητήσεις ε, δεν είναι γνωστές. Και δεν θα ξέρουμε πολύ σύντομα αν θα πετύχει, εν πάση περιπτώσει, κάτι περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκτώντας χώρο για κίνηση, περισσότερο από όσο έχει. Ρυθμέρκης, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έτσι γρήγορα. Συζητήσαμε το ότι πετάμε όλο και περισσότερο. Εγώ θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών είναι καλό σύστημα. Καλό είναι να μην το αντικαταστήσουμε γιατί και το νέο σύστημα θα έχει παιδικές αρρώστιες δεν υπάρχει επαρκή πίεση στον ΑΙΚΑΟ αυτή τη στιγμή για να φέρει ένα νέο σύστημα φέτος, κάτι το οποίο χρειάζεται. Δεν θεωρώ πως η λύση πρέπει να είναι να μην περιοριστεί η αεροπορία. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι για να παραμείνει εντός των φιλοδοξιών της, εντός του συστήματος και να δώσει χώρο στην αεροπορικό τομέα να παραμείνει κερδοφόρος. Δεν θεωρώ πως θα αντικατασταθεί το σύστημα αυτό με κάποιο άλλο. Είναι δύσκολο να αντικατασταθούν αυτά τα αισθήματα. Δεν βλέπω εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, ένα νέο σύστημα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα ήθελα. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν τώρα αν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ποιο, θα πάρει το λόγο από σας. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής που έχουν λάβει το λόγο για την προτινόμενη εξαίρεση. Θα παραμείνω τώρα στο επίπεδο της συνοπτικότητος σε ό,τι αφορά την ε, επέκταση του σφαίρα εφαρμογής για να καλύψουμε και πτήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να θυμηθείτε από πού προέκυψε αυτό. Αυτό ήταν ε, αντιμετώπιση μιας δυναμικής που είχε αντιμετωπιση μιας δυναμικη που μέσα στην ΙΚΑΟ για να προετοιμαστεί το έδαφος διαπραγματεύσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με το σύστημα ETS για τους Ελβετούς εταίρους μας. Η κατάσταση δεν ήταν ακριβώς η ίδια. Οι Ελβετοί δεν έχουν ποτέ διαμφισβητήσει το σύστημα ETS και είναι σε διαπραγματεύσεις θέλοντας να συνδέσουν το ελβετικό σύστημα με το ευρωπαϊκό σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών. Αυτό δημιουργεί ειδικέ συνθήκες που είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της γεωγραφικής θέσεις της ε, Ελβετίας που είναι στη μέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους κοινού στόχους και την ιδεολογική συγγένεια των Ελβετών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε λοιπόν ότι το να παρατείνουμε αυτή την εξαίρεση δεν πρόκειται να βοηθήσει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το κόστος και τις πιθανές στρεβλώσεις ανταγωνισμού, όλοι οι φορείς που κάνουν πτήσεις μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, κάποιες ε, αεροπορικές εταιρείες έχουν υπολογίσει το κόστος 25 cents για κάθε πτήση αυτό, και κάθε επιβάτη. Αυτό δεν πρόκειται λοιπόν να αλλάξει τα σχέδια διακοπών κανενός. Τέλος, σε σχέση με τις διεθνείς ε, πιστώσει στον τομέα αυτό. Εμείς έχουμε σχεδιάσει τις ε, εξαιρέσεις μας με έναν τρόπο που είναι μινιμαλιστικό και διατηρεί και την ακαιρεότητα και τα αρχικά σχέδια του ETS και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει μια αξιόπιστη εξαίρεση για ένα χρόνο. Θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην εφαρμογή του συστήματος ε, ETS πλήρως σε ένα χρόνο εάν δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία. Δεν έχουμε αλλάξει τα ποσοστά σε σχέση με το, την διεθνή αυτή υποχρέωση παραμένει στο 15%. Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν αγοράσει αυτές τις, ε, αυτά τα δικαιώματα για οικουμενική κάλυψη θα μείνουν με κάποια πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια και θα μπορέσουν να τα πουλήσουν και αυτά στην διεθνή αγορά. Όταν γίνονται λοιπόν έκτακτες αλλαγές θα προκύπτουν και έκτακτες συνέπειες. Αλλά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την εξαίρεση είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία πολύ περισσότερα από τις ζημίες που θα προκύπταν από μια πλήρη αγορά των διεθνών ε, πιστώσεων. Πρέπει να το δούμε αυτό λοιπόν σε συνολικό πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο Πέτερ Λίζε ο συζητητής, για να κλείσει τη συζήτηση πάρα πολύ σύντομα. Αυτοί οι οποίοι <clears throat> υποστήριξαν τις θέσεις μου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αντιμετωπίσω. Ο Μάρτιν Κάλενεν αντιμετώπισε και πάλι το θέμα των εσόδων του, τι θα κάνουμε με αυτά. Βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αν υπάρξει μια τροπολογία λοιπόν για τον προσδιορισμό για το earmarking θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα κονδύλια και υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυσκολίες με τα τρίτη, τρίτα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν είπε ότι ούτως ή άλλως μέχρι τον Απρίλιο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, δεν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, αλλά δεν θα είναι ιδιαίτερα θετικό εμείς ως νομοθέτες να μην καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ή λοιπόν θα υπάρξει μια συμφωνία, αλλιώ θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι η συμφωνία. Από την άλλη πλευρά όμω, ο Μάτιν και ο Κρίς θα πρέπει να ξέρουν ότι κάτι έχει αλλάξει από το 2008 μέχρι τώρα. Το 2008 δεν είχαμε κατανοήσει πόσο μεγάλη είναι η αντίδραση των κρατών ε, μελών των τρίτων κρατών. Και δεν πρέπει αυτό να μα οδηγήσει στο να εγκαταλείψουμε την κλιματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επικοδομητικέ ενέργειε. Νομίζω ότι με του Αμερικανού <clears throat> υπάρχει ένα κοινό συμφέρον και πρέπει να καταλήξουμε σε κοινέ προσπάθειε για να δούμε πώ θα γίνει η χρηματοδότηση αυτών των, ε, η χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων και σίγουρα είναι μια θετική πρόταση προς τα αναπτυσσόμενα κράτη όταν τους λέμε ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη. Και για μένα το είπαν πολλοί ότι είναι πιο σημαντική η χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων από το να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε για τα θέματα αυτά και θα πρέπει ως το Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση και όχι να πετάμε το φταίξιμο ο ένας στον άλλο. Ο Καρσουίτερ είπε δεν χρειάζεται να σταματήσει το ρολόι, Δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατό. <clears throat> Αν θέλουμε να έχουμε μια διεθνή συμφωνία θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαδικασία. Η Φρανσουάς Κοστέτ είπε κάτι, έκανε μια τροπολογία που είναι πάρα πολύ τεχνικού χαρακτήρα. Πρέπει να δω ακριβώς τι λέει το αρχικό γαλλικό κείμενο. Ο Γκακράμερ μίλησε για το πρόβλημα με την ε, Ελβετία που είναι ευαίσθητο θέμα και η Κομισιόν ίσως δεν έχει δράσει με τον πιο διπλωματικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η επίκρισή μας εναντίον της Κομισιόν. Γιατί η Ελβετία δεν έχει ποτέ επικρίνει το σύστημά μας, πάντα ήταν στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς θα ήταν πιο ευφυές να λάβουμε υπόψη τα επιχειρήματα της Ελβετίας. Και τέλος υπάρχει το θέμα του να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι η Ελβετία θα καταφύγει στα δικαστήρια έναντι αυτής της ε, απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το να έχουμε πτήσεις από την Ζηρίχη που να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως οι πτήσεις από το Μόναχο ή οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιες αντιδράσεις από την πλευρά των Ελβετών. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια σωστή ρύθμιση η οποία θα είναι νομικά ε, στεγανή. Μια σωστή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση που θα συμπεριλάβει και την Ελβετία το παράδειγμα με το Düsseldorf και τις πτήσεις από τη Μαγιόρκα στην Αίπτο είναι ίσως το πιο λαθασμένο παράδειγμα. Η Κομισιόν έχει αναφέρει εταιρείε που πετούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συμπεριλάβει στα, στους ναύλους τους το κόστος του ETS, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόστος αυτό. Αυτή τη στιγμή ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλό, ούτε 25 cents και ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αλλάξει την καταναλωτική συμπεριφορά κανενός ένα, μια επιβάρυνση 25 cents. Για αυτά λοιπόν τα οποία ισχύουν τώρα το 2012 έχουμε ήδη ένα επίπεδο κυρώσεων το οποίο δεν είναι επαρκέ για να αλλάξει συμπεριφορά και θα ήταν παράλογο να πιστεύει κανεί ότι θα προτιμήσει να πάει στην Αίγυπτο από τη Μαγιόρκα αντί να πάει στη Μαγιόρκα από τον Ντίσσελντοφ επειδή είναι η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση από το ETS. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτά τα επιχειρήματα και να εστιάσουμε στην επίτευξη διεθνούς συμφωνία. Πιστεύω ότι ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να αποφασίσει εάν τον επηρεάζουν όλα αυτά ή όχι. 26 Φεβρουαρίου θα αποφασίσουμε στην Επιτροπή ε, επί, ε, περιβάλλοντος και τον Απρίλιο ελπίζουμε ότι θα συζητήσουμε για τη διαδικασία σταματήματος του ορολογίου. Ερχόμαστε τώρα στο ήπιο κρέας που είναι το επόμενο θέμα, ένα καυτό ζήτημα και έχω πάρει πολλές ε, αιτήσει στο θέμα αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη και φυσικά θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αιτήσει. να δούμε ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Είχαμε ήδη το 2011 το θέμα αυτό στην ημέρησια διάταξη της Επιτροπής μας, αλλά δεν προήλθανε από τη συζήτηση αυτή οι ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα και καλύτερη ετικετοθεσία. Εγώ θέλω τώρα να χαιρετήσω την παρουσία του Συμβουλίου και της κυρίας Τεστόρη από την ε, ε, Γενική Διευθυνσή ΣΑΝΚΟ Ξέρουμε ότι υπάρχει μια εργόδης τώρα δραστηριότητα για τα θέματα αυτά, εθνικά σχέδια τα οποία είναι υπό επεξεργασία. Όλα αυτά μας κάνουν να κατανοούμε ότι χρειάζεται μια καλύτερη ευρωπαϊκή ρύθμιση, μια πιο στεναρή ρύθμιση και επομένως θα δώσω το λόγο στους συντονιστές καταρχήν και μετά στους επόμενους, στους υπόλοιπους συναδέρφους. Θα μαζέψουμε τις παρεμβάσεις για να δώσουμε το λόγο μετά στο Συμβούλιο και θα ήθελα σε όλους να ζητήσω να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι σύντομοι ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Και ξεκινώ με τον Πέτερ Λίζε για το ΕΛΚ και μετά η Λίντα Μακ Ιουαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ πέρα με τη λανθασμένη σήμανση του κρέατος του αλογίσιου που σημαίνει ως ε, βόηο είναι μια ε, απάτη και αντιλαμβάνομαι τον ε, κάθε καταναλωτή που λέει εγώ δεν θέλω να φάω άλογο. Και κατανοητές και αντιδράσεις. Τώρα, είμαι κάπως επιφυλακτικός για την απέτηση για τη σήμανση της προέλευσης όλων των πιθανών συστατικών. Και θα ήθελα να μου πει κάποιος εδώ πέρα από την αίθουσα το αν έγραφε πάνω βόλιο κρέας προέλευση Ρουμανία ή προέλευση Γαλλία αντί για βόλιο κρέας σε τι θα βοηθούσε. Το πρόβλημα ήταν πως είχε κρέας αλόγου και έγραφε πάνω βόλιο. Αυτό ε, δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία, χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης. Γι' αυτό χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν αυξάνει τους ελέγχους, θα κάνει τεστ ε, DNA και χαίρομαι που είναι εδώ πέρα και η κυρία Τεστόρη. Θα ήμουν ε, κάπως αμήχανος να ασκήσω κριτική στον ε, κύριο Μπόργκ γιατί δεν φταίει και για την πολιτική της Κομισιόν μέχρι τώρα. Υπενθυμίζω εδώ πέρα στη Λίντα Μακάβαν, Πιλάρα Γιούζο κτλ που ήταν παρούσες όταν πριν από λίγα χρόνια ζήτησε το Κοινοβούλιο ε, την ε, σήμανση της δεύτερης και τρίτης γενιάς ε, του κρέατος από και είχε πει η Κομισιόν πως δεν μπορεί να το ελέγξει. Επειδή όμως εγώ γνωρίζω τα, τα της γενετικής είπα κάντε ένα τεστ DNA. Και όπως είπα αντιλαμβάνομαι την οργή του καταναλωτικού κενού. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα της προστασίας των ζώων γιατί εδώ πέρα είναι ακόμη πιο σημαντική υπόθεση ο κλονισμός και υπάρχουν σοβαρές ε, ανησυχίες στον τομέα της υγείας κτλ. Ε, και επίσης και με τα κατάλοιπα των ε, φαρμάκων είναι σοβαρό το ζήτημα, αλλά με το, με το κρέας από κλόνους έχει ακόμη περισσότερο λόγο να πει ο καταναλωτής θέλω να ξέρω τι τρώω. Και άμα μου λέτε ότι κοστίζει το κρέας το τεστ με συγχωρείτε DNA δεν είναι δυνατόν να ζητάμε κάτι και να μας λέτε πως ε, δεν γίνεται η Κομισιόν πρέπει γρήγορα να υποβάλει πρόταση για το, για το κρέας από Και θα ήθελα εδώ πέρα να μας πείτε συγκεκριμένα το τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ, Λίντα Μακάβανη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που σώκαρε σχετικά με το κρέας από άλογο είναι ότι το σύστημα ανιχνευσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέτυχε. Και δεν υπάρχει από το σφαγείο και μετά. Και το τι ακριβώς κρέας μπαίνει στο ψιλοκομμένο κρέας, τον κοιμά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζει κανείς. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της ετικετοθεσίας και της σήμανσης ε, ε, των προϊόντων. Κάποιες προτάσεις που είχαν γίνει, πολλοί συνάδελφοι τις απέρριψαν και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Και να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε γύρω από το θέμα αυτό. Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, έγιναν κάποιες προτάσεις θα το συζητήσουν επιτέλους. Θα είμαι σύντομη πάντως γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι που φέρουν το λόγο. Πριν λίγο χρόνια είχαμε μία συζήτηση για την υγιεινή της παραγωγής, της διαδικασίας παραγωγής κρέατος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την εντύπωση ότι θέλει να εξασθενήσει κάποιες, ε, κάποιους κανόνες, δεν θέλει να υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεγκτές στα σφαγεία και αυτό είναι, κρίθηκε αρνητικό από μας. Μετά από όλα αυτά που είδαμε ότι συμβαίνουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ε, πιστεύετε ότι το κοινό θα δεχθεί οι επιχειρήσεις να είναι υπεύθυνε μόνες τους για τον έλεγχο της παραγωγής τους ή μήπως θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει η Επιτροπή να κρατήσει το σύστημα των ανεξαρτήτων ελεγκτών. Υπάρχει πίεση από ό,τι φαίνεται και από τις επιχειρήσεις, υπάρχει πίεση και από τις κυβερνήσεις. Τι ακριβώς θέλει να κάνει η Επιτροπή, θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι πλέον λύση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων τόσες φορές στην Επιτροπή μας. Αλλά αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα όταν ο καταναλωτής αγοράζει κάτι το οποίο λέει ότι είναι βόλιο κρέας και είναι αλογίσιο. Θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι καταρχήν μια εθνική υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα κάθε κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι το κρέα που πωλείται σε μια χώρα ακολουθεί την νομοθεσία. Το λέω αυτό γιατί είναι ο κύριο Πολ εδώ πέρα. Είναι πολύ ε, Σπάνια η παρουσία, τόσο σπάνια όσο ένας γνήσιος, ένα γνήσιο μπιφτέκι από βόλιο κρέας. <clears throat> Αλλά υπάρχουν χώρες όπου είναι αποδεκτό το να τρώει κανείς ε, αλογίσιο κρέας. Φανταστείτε να έχουμε κρέας που περιείχε χείριο κρέας που θα είχαμε τεράστια προβλήματα από τις θρησκευτικέ κοινότητες στην Ευρώπη θα θεωρεί το η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα επιλήψιμος. Μπορείτε να καταλάβετε πώς οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι θα αντιμετωπίζανε κάτι τέτοιο. Η ευθύνη λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο των παραγωγών τροφίμων. Αυτοί αγοράζουν τα, το κρέας, αυτοί αγοράζουν τα προϊόντα αυτά αυτοί βάζουν την τελική σφραγίδα για τα τρόφιμα, επομένω αυτοί έχουν την ευθύνη για την σωστή ετικετοθεσία και σήμανση των προϊόντων αυτών. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που απαιτεί να υπάρχει αυτή η σήμανση, αλλά αυτό εξαρτάται από τι εθνικέ κυβερνήσει που θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία με έναν τρόπο ο οποίο είναι αποτελεσματικό, είναι αναλογικό και είναι αποτρεπτικό για αυτού που θέλουν να κάνουν απάτε. Έχουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Έχουμε κάτι τέτοιο που να δείχνει ότι εφαρμόζεται ο νόμος, ότι υπάρχουν παραγωγός χάρη κυρώσεις για λανθασμένη ή απατηλή σήμανση, ότι οι κυρώσεις αυτές έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα, υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ του τρόπου εφαρμογής αυτού του νόμου μεταξύ διαφορών χωρών και πώς τα δικαστήρια θα αντιμετωπίσουν αυτή την νομοθεσία. Εγώ δεν είδα κάποιον να λέει ότι δεν τολμούμε να κάνουμε τους σωστούς ελέγχους από τους παραγωγούς τροφίμων, γιατί άμα κάνουμε αυτές τις ε, δοκιμασίες θα μας απαγορεύσουν να παράγουμε τρόφιμα. Εγώ ξέρω μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε άλλες χώρες, αλλά ξέρω ότι στην χώρα μου αυτό έχει αντιμετωπιστεί σαν ένα πραγματικά αποτρόπαιο αδίκημα. Θέλουμε να έχουμε μια ενιαία αγορά, θέλουμε τα τρόφιμα να περνούν από τη μια χώρα στην άλλη, θέλουμε να οι κυρώσει. Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να γίνονται κάποιε προσπάθειε να εναρμονίσουμε τι κυρώσει ώστε να είναι πραγματικά αποτρεπτικέ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πολλοί από εμά δεν θέλουν να το κάνουν καν. Αλλά τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να έρθει στην προσοχή των κρατών μελών, να κάνουμε συγκρίσει για τι κυρώσει που επιβάλλονται μεταξύ κρατών μελών. Και το ερώτημα είναι πώ μια χώρα επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ και μια άλλη χώρα λέει ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές διώξεις λόγω αυτού. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας εξηγήσει τι είδους μελέτες κάνει, τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το αποτελεσματικός, αναλογικός και αποτρεπτικός, αυτά τα τρία επίθετα μπορούν να ισχύουν στα κάτι μέλη. Ε, ευχαριστώ. Ο Κάρλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε συζητήσει το θέμα της σήμανσης ε, των τροφίμων και ένας από τους ε, λόγους γιατί θα βοηθούσε η ετικέτα, η σήμανση αυτή, είναι ότι ε, υπάρχει η δυνατότητα να διευκρινίζεται η αναζήτηση του ευθυνότερου κάθε φορά παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαμεσολάβηση εμπόρων, διαδοχικής αλυσίδας εμπόρων που στην ουσία οδηγούν στην αύξηση της τιμής παρά την αναζήτηση της φθηνότερης τιμής παραγωγής. Αν έχεις μια πιο μόνιμη σχέση με τους παραγωγούς θα είναι δύσκολο να αλλάξεις και θα είναι δύσκολο να αλλάζεις συνεχώς και τη σήμανση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί λοιπόν η καταγωγή και η προέλευση μάλλον των κρεάτων όπως επίσης το βλέπουμε ότι είναι δύσκολο και στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων. Και όπως έχουμε πει σήμερα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο το να κάνει κανείς τέτοιου είδους λάθη. Πριν δύο χρόνια η αρμόδια υπηρεσία στη Σουηδία εξέτασε ε, τις ετικέτες. 44% ήταν ε, λανθασμένες οι ετικέτες. 70% των έτοιμων φαγητών ήταν επίσης ε, λανθασμένη η ετικετοθεσία τους. Τίποτα δεν έγινε, κανένας δεν τιμωρήθηκε. Δεν ελήφθη καμία κύρωση εις βάρος όλων αυτών. Ο κίνδυνος λοιπόν ε, για την ανακάλυψη μιας ε, απάτης είναι πάρα πολύ μικρός. Ε, πολλές φορές η αναζήτηση του κέρδους με παράνομο τρόπο είναι τρομακτικό κίνητρο. Το να συγκεντρώνει κανείς την προσοχή του αποκλειστικά στο φινότερο σημείο παραγωγής, αυτό είναι κάτι δυστυχώς που αυξάνει τις πιθανότητες απάτης. Πρέπει να αλλάξει μια τέτοια λογική. Και κυρίως ε, όταν κάποιος κάνει κάτι το απαράδεκτο πρέπει να το νιώθει η επιχείρηση, να υπάρχουν κυρώσεις εις βάρος της. Οι αρχές ελέγχου βλέπουν τις επιχειρήσεις σαν συνεταίρους σχεδόν, σαν φίλους και όχι ε, σαν ε, ελεγχόμενα, σαν ελεγχόμενες οντότητες. Φυσικά πρέπει να έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά όταν μια επιχείρηση κάνει κάτι το άσχημο, θα πρέπει να επιβάλλεται ένα πρόστιμο και όπου υπάρχει εγκληματική απάτη, ακόμα και φυλάκιση των υπευθύνων. Chris ε, Davis, ε, δεν είναι πρώτη φορά που ξέρουμε ότι ένα λάθος προϊόν βρίσκεται σε άλλο, στη θέση κάποιο άλλο. Ε, έχει συμβεί και στο παρελθόν και στη Σουηδία πέρυσι είχαμε χείριο κρέας με ετικέτα βόλιο και είχαν προσθέσει χρώματα για να φαίνεται σαν βόλιο και κανένας ε, δεν το, δεν σχολίασε εκτός αν οι πελάτε, όταν οι πελάτες είπαν ότι αυτό δεν έχει γεύση εν πάση περιπτώσει βοήου κρέατος και τότε ε, ανακαλύφθηκαν οι απάντες. Λοιπόν, τα συστήματα ελέγχου τα οποία έχουμε κανονικά θα έπρεπε να τα ανακαλύψουν όλα αυτά και η ΕΦΣΑ και οι, τοπι, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί μέχρι τώρα απέτυχαν. Εμείς έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε ε, το φινότε, τη φινότερη τιμή για τα τρόφιμά μας και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πρότυπα ποιότητας υψηλά. Θα πρέπει να συνηθίσουμε ε, ότι στο μέλλον τα τρόφιμα θα πάρουν μεγαλύτερο τμήμα των ισοδυνάτων μας εκτός και αν στρέψουμε την προσοχή μας στην ποιότητα γιατί όταν συγκεντρωνόμεθα αποκλειστικά στο ευθυνότερο της τιμής ε, του κάθε τέτοιου προϊόντος τότε θα έχουμε απάτες σαν τη σημερινή όλο και πιο συχνές. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν ο πολιτισμός της διατροφής. Θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να υπάρξει καλύτερη συνεργασία, να υπάρχουν ε, ισχυρές κυρώσεις αν κάποιος κάνει ε, παράνομες ενέργειες και θα πρέπει να σεβαστούμε τους καταναλωτές, θα πρέπει να σεβαστούμε την ευημερία των ζώων και οι καταναλωτές που έχουν ανάγκη ε, φθηνά τρόφιμα να τρώνε λιγότερο κρέας ή σε μικρότερες ε, μερίδες. Ε, όταν ήμουν παιδί τρώγαμε πολύ λιγότερο κρέας από ό,τι σήμερα και είχαμε ε, με την ίδια τιμή ε, περισσότερα λαχανικά, προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε το περιβάλλον και εκτιθέμεθα λιγότερο σε κινδύνους τρώγοντας λιγότερο κρέας και έτσι μειώνουμε και την πιθανότητα να μας εξαπατήσει η βιομηχανία. Ροσμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν και βεβαίως για μένα σε κάποιες χώρες της Ευρώπη είχαμε παράδοση υψηρά να τρώμε κρέας αλόγου. Οπότε για μένα δεν είναι ζήτημα διατροφικής ασφάλειας, αλλά ζήτημα ίχνη λασιμότητας και σήμανσης. Και απάτη επίσης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Αλλά αν εγώ έχω μια εταιρεία και παρακολουκάνικα, θα ήθελα να έχω την ίδια ποιότητα κάθε εβδομάδα. Οπότε θα πρέπει να ξέρω τι ακριβώς βάζω σε αυτά τα λουκάνικα. Μέχρι κεραίας. Για να έχω κάθε ε, εβδομάδα την ε, ίδια παραγωγή. Οπότε δεν είναι θέμα σήμανσης. Είναι ζήτημα του να θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Επίσης, από πού προέρχεται το κρέας. Άμα μιλάμε για Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Από πού και να προέρχεται. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα σταματήσει η ανεντιμότητα και πώς θα τιμωρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω πρόβλημα με το κρέας του αλόγου, απλά το πώς έγινε. Και περισσότερο νομίζω δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς οι εταιρείε θα καταλάβουν πώς πρέπει να πουλάνε σωστό κρέας και πως όλοι έχουν δικαίωμα να ξέρουν από πού προέρχεται το φαγητό τους ε, για να πούν δεν θέλω να αγοράσω αυτό το προϊόν ή θέλω να το αγοράσω. Και ε, νομίζω πως το σύστημα εδώ είναι μεγάλο και πρέπει να ε, σκεφτούμε ένα πακέτο μέτρων και όχι μόνο να πούμε πως είμαστε κατά και δεν θέλουμε να ξαναγίνει. Πρέπει να είμαστε και εμείς δημιουργικοί, να βρούμε ένα σωστό πακέτο για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με πολλούς προλαλήσαντες. Πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής τι έχουν μέσα τα φαγητά του και πολλές φορές έχουμε συζητήσει εδώ πέρα το πώς μπορούμε καλύτερα να σημάνουμε τα τρόφιμα και να σημαίνουμε τα τρόφιμα και επίσης τα της ε, προέλευσης. Επρόκειτο λοιπόν για έναν ε, Ολλανδό, ο οποίος ε, είχε μια εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, σφάχτηκαν τα ζώα, όπως ξέρετε, στη Ρουμανία, πήγαν σε μια γαλλική εταιρεία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά κάπου σε ολόκληρη αυτή την ε, αλυσίδα μπήκε μια ετικέτα βόηου κρέατος ε, αλογίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσει πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατόπιν σταμάτησε η παραγωγή του ε, παρασκευαστηρίου αυτού στην ε, Ολλανδία και εκεί πέρα ανακατεύθηκαν τα δύο κρέατα παρά το ότι υπήρχε η ετικέτα ότι ήταν 100% βόλιο κρέας. Είναι σαφές πως πολλές εταιρείε στην ε, Ολλανδία αλλά και αλλού δεν εφαρμόζουν καλά τους ε, κανόνες και άρα μετά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει τι βρίσκεται μέσα στο χάμπουργκερ του. Ζητάω λοιπόν από την Κομισιό να κάνει κάτι και να κινηθεί ειδικά κατά αυτών των κρατών που παραβίασαν την σχετική νομοθεσία. Επίσης ε, βλέπω πως ε, όταν μιλάμε για τα καινοτόμα λεγόμενα τρόφιμα, δηλαδή για τα το κρέας από κλόνους. Ε, μας έλεγε η Κομισιόν ε, πως ε, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το οποίο ζητάμε, δηλαδή τεστ DNA, αλλά τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μπόρκ μας είπε πως θα γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει με την εχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών και ειδικά όταν μιλάμε για το βοδινό κρέας. Εκ πρώτη όψεω μοιάζει να είναι μόνο ζήτημα λάθος ε, σήμανση. αλλά σιγά σιγά εξελίσσεται σε ζήτημα διατροφικής ασφαλείας. γιατί από ό,τι φαίνεται πως ε, τα άλογα, φαίνεται πως τα άλογα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν εισαχθεί ποτέ στη διατροφική αλυσίδα. Δεν ξέρουμε τι φάρμακα είχαν πάρει και υπάρχει πιθανός ε, κίνδυνος υγείας και θέλω να μας πει η ΕΦΣΑ τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Και η Κομισιόν τη σκοπεύει να κάνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολ Νούτελ. Σας καλωσορίζω στην ε, Επιτροπή μας. Είναι πρεμιέρα σήμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ευχαριστώ τον συνάδελφό μου και τον Chris Davis που παρατηρήσε την παρουσία μου. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως ο Βρετανικός τύπος έχει αγνοήσει το, την πτυχή την ευρωπαϊκή για το σκάνδαλο αυτό γιατί ε, ειλικρινά τα τρία πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε είναι τα εξή: ε, Η διατροφική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 178 του 2002 με τον οποίο η αρμοδιότητα πήγε από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες και υπάρχει και 854 του 2004. Πριν από αυτούς τους κανονισμούς είχαμε πολύ ε, αυστηρές προδιαγραφές στον Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της ε, κρίσης ε, της φογκόδους εγκεφαλοπάθειας. Και αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πως ε, μετακύλησε την ευθύνη στους παραγωγούς αντί στις ε, αρμόδιες αρχές. Ο Chris Davis είπε πως ευθύνονται και τα κράτη-μέλη. Ας δούμε την οδηγία 2000 κάθτος 13 κάθτος ΕΚ. Μπροστά μου την έχω. Η σήμανση ξεκάθαρα είναι και αυτή αρμοδιότητα της Ένωσης. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν διασφαλίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων και το σημαίνουμε και λάθος. Ο κόσμος τρώει άλλο κρέας από αυτό που νομίζει ότι αγόρασε και σε κάποιες περιπτώσεις α, υπάρχει κόσμος που φύγεται από το άλογο. Εμένα μου αρέσει, εντάξει, αλλά κάποιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να το ανεχτούν. Το τρίτο πρόβλημα που βλέπω είναι η πολύ αγαπημένη μας ε, ενιαία αγορά που τόσο μας εμπνέει. Λες και θα κατέρεε ο κόσμος εάν βγαίναμε από την ενιαία αγορά. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις το κρέας έχει ταξιδέψει σε πέντε χώρες. Σε πέντε χώρες η διατροφική αλυσίδα. Εγώ θεωρώ πως είναι αδύνατον να ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και διασφαλίζει η ιστορική ε, αγορά πως ε, τα σύνορα διασχίζονται με ελάχιστο έλεγχο. Εγώ θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να επανέλθουν στα κράτη-μέλη αυτές οι αρμοδιότητες γιατί θεωρώ πως ε, μπορούμε να μειώσουμε έτσι τη γραφειοκρατία, μπορούμε να γίνουμε ακόμη πιο αυτάρκης και να μην βασιζόμαστε σε άλλες χώρες και οι καταναλωτές θα είναι πιο προστατευμένοι. Και αυτό το οποίο ελπίζω και πραγματικά δεν θέλω να το κάνει η Κομισιόν είναι να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση για να αυξήσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τι συμβαίνει. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είτε στον οικονομικό τομέα, είτε στον τομέα των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση το εκμεταλλεύεται για να αρπάξει ακόμη περισσότερη εξουσία στις Βρυξέλλες και να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τις εθνικές δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν για τα λόγια σας. Και περνάμε τώρα στους άλλους ομιλητές. Σας λέω τον κατάλογο. 1,5 λεπτό ο καθένας για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Η κυρία Γκροστέτ. Der Kollege Gerbrandi,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 Και κλείνω με τον ομιλητή αυτό το κατάλογο. 1,5 λεπτό λοιπόν για όλους. Παρακαλώ να παραμείνετε σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν όλοι να έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσει. Φρανσουάζ Ντροστέτ, σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μια απάτη. Το πρόβλημα είναι ότι ο κάθε κρίκος της αλυσίδας κάνει πάσα το φταίξιμο στον άλλο. Μέσα στα πλαίσια της ενίας αγοράς υπάρχουν όλο και περισσότερο στάδια και κρίκη στην αλυσίδα και ο έλεγχος είναι όλο και πιο δύσκολος. Και ιδίω όταν πρόκειται για απάτη για μεταποιημένα τρόφιμα. Όταν φανταστούμε το πόσοι τόνοι χρειάζονται για να φτάσουμε σε αυτά τα προϊόντα, δεν καταλαβαίνω. Ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανάμειξη πρώτων υλών που προέρχονται από πάρα πολλές προελεύσεις. Το ερώτημά μου είναι μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους κρίκους με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε την εχνηλασιμότητα για τα μεταποιημένα τρόφιμα. Επίσης τα τεστ DNA που πρέπει να γίνουν για τα προϊόντα που έχουν ετικετοθεσία βοδινό. Πόσο θα κοστίσουν αυτά πώς θα μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των δοκιμασιών που θα γίνουν και επί ποιας βάση. Πώς θα έχουμε ένα ε, αντιπροσωπευτικό δείγμα. Πώς θα έχουμε λοιπόν μία... Γιατί να μην είναι μονάχα μια σύσταση και γιατί να θέλουμε να κάνουμε υποχρεωτική αυτή η δοκιμασία. Είναι απαραίτητο να έχουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και έχουμε πολλά να κάνουμε. Η Όσα Βέσλοντ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά έχουν ελεγχθεί ήδη για μένα όμως είναι πάρα πολύ σαφές ότι οποιοδήποτε ο οποίος ισχυρίζεται ότι το κρέας αυτό είναι βόηο, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι είναι βόηο το κρέας. Οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν που πούλησαν αυτά τα προϊόντα με το φτηνό αυτό κρέας για να βγάλουν λεφτά, δεν έχουν επομιστεί τις ευθύνες τους να το ελέγξουν προτού το πωλήσουν στους καταναλωτές. Μετά από το σκάνδαλο λοιπόν <clears throat> και πάλι δεν έχουν κάνει αρκετά. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει η κοινωνία για να αυξήσει τους ελέγχους. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα προς την Κομισιόν. Να το κάνω όμως πιο στενάρο το ερώτημα αυτό. Τι θα κάνετε για να ενισχύσετε τους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Πώς θα σχεδιάσετε τους ελέγχους αυτούς σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να εξασφαλίσετε ότι υπάρχουν κριτήρια ασφάλειας και ώστε να εξασφαλίσετε ότι μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια των ετικετών και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις για τους παραγωγούς τροφίμων και τους εμπόρους τροφίμων αν υπάρχουν προβλήματα. Ξέρω ότι για την, ε, ε, για την περί προέλευσης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό θα αναγκάσει τις εταιρείε να ελέγχουν από πού έρχεται το κρέας τους και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα. Θα είναι πιο ισχυρό λοιπόν το στοιχείο αυτό. Η Πίλαρ Αϊούσο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία. Είναι σαφές ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία απάτη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις προδιαγραφές που ισχύουν για αυτά. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η κύρωση. Στη χώρα μου έχουμε ένα νόμο περί απατών που καθορίζει το πρόστιμο σαν συνάρτηση του κέρδους που προήλθε από αυτή την απάτη. Και έχουν τεθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα για περιπτώσεις απατών που δεν ήταν τροφιμικού χαρακτήρα. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω στην Κομισιόν είναι το εξής. Φαίνεται ότι βρέθηκε φενιλβουτασόνη σε αυτό το κρέας αλόγου που μπήκε στην τροφιμική αλυσίδα. Αυτή η φενιλοβουτασόνη χρησιμοποιείται για τα άλογα κούρσας, όχι για τα άλογα τα οποία το κρέας θα καταναλωθεί. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόνα μου που, πού βρέθηκε αυτή η ουσία, γιατί αυτό πράγματι θέτει ένα πρόβλημα τροφιμικής ασφάλειας. Ευχαριστώ, Ελένη Σβίγματ. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι οι υπουργοί κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ετοκρισία, ενώ το 2011 είχα καταθέσει τροπολογίες που δεν υποστηρίχθηκαν από το έλκα, αλλά έγιναν δεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υποστηρίχθηκαν από το Συμβούλιο και δεν έγινε τίποτα με αυτές τις συστάσεις. Λοιπόν, καταλήξαμε απλά σε μια έκθεση χωρίς συνέχεια. Δεν έχουμε κάνει ρυθμίσεις για επεξεργασμένα τρόφιμα, για το κρέα στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα κρέατα προέρχονται από 13 διαφορετικές προελεύσεις. Θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής από πού προέρχονται όλα αυτά και αν είναι η ετικετοθεσία λανθασμένη αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ξαφνικά δυστυχώς όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε δεν ισχύουν για τα επεξεργασμένα τρόφιμα και μάλιστα σε κάποια έτοιμα τρόφιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν και ίχνη από χείριο κρέας. Πρέπει λοιπόν οι προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε να είναι αυστηρές και να προχωρήσουν με μεγάλη ταχύτητα για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όταν ο κόσμος αγοράζει βόλιο κρέας δεν ξέρει αν είναι βόλιο ή είναι από άλογο, αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Μακίνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ιρλανδία το ανακάλυψε γιατί έψαχνε και νομίζω πως είναι ένα καλό παράδειγμα του τι πρέπει να κάνει μια υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων. Και καλό είναι να ακούσουμε κάποια στιγμή τον ε, διευθυντή, τον κύριο Άλαν Ράιλι, που είχε ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Δύο μηνύματα. Πρώτον, το να ασχολούμαστε με τη σήμανση είναι λάθος, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για μια απάτη. Και οι εγκληματίες ε, δεν το δηλώνουν στην ετικέτα. Ε, η ετικέτα μπαίνει στα πάντα. εάν δεν δούμε τι υπάρχει μέσα στο κουτί, τότε δεν έχει καμία αξία η ετικέτα. Στην Ιλλανδία ανακαλύψαμε πως ε, αυτό το οποίο είχε πάνω ετικέτα ε, βόλιο κρέας ήταν ε, άλογο και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτή την αρχή. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που θέλει ευρωπαϊκή λύση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, έχουμε πολύ αυστηρή ίχνη λασιμότητα των ε, βοδινών. Χρειαζόμαστε καλύτερη ίχνη λασιμότητα και για το κρέας αλογού. Και θέλω να μας πει η Κομισιόν πώς θα γίνει αυτό. Πόσο, ε, σε ποιο βαθμό υπάρχει λασιμότητα. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε πιο αυστηρούς κανόνες για τα άλογα, εάν μπουν στην τροφική αλυσίδα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα πέρα από το ζήτημα της ευζωίας. Και επειδή ε, το ανακάλυψε η Ιρλανδία, θα ξεπεράσω λίγο και το χρόνο μου κύριε Πρόεδρε για το θέμα της συχνασιμότητας. Πρέπει να το πω. Ο Καρλ το είπε. Ε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Κάθε συνάδελφος θέλει να μιλήσει. 1,5 λεπτό. Λοιπόν, Κόριν Λεπάζ. Ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Έχουμε το αποτελέσματα ενός συστήματος μέσα στο οποίο κάθε φορά που επιθυνούμε κάποιοι από εμά να υπάρξει μια υποχρεωτική δεσμευτική ρύθμιση, στην ουσία μας οδηγούν πάντα σε ρυθμίσεις οι οποίες είναι εθελοντικές. Όταν ζητάμε αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας λένε ότι τα κράτη πρέπει να το κάνουν. Τα κράτη για οικονομικούς λόγους κάνουν όλο και λιγότερους και το σύστημα καταλήγει στο να μην δουλεύει. Εάν πράγματι θέλουμε εμείς οι συμπολίτε μας να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στα προϊόντα που καταναλώνουν, πρέπει να υπάρχει σωστή ετοκιτοθεσία για την προέλευση του κρέατος, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ακόμα και στα προπαρασκευασμένα γεύματα από πού προέρχεται το κρέας. Το σύστημα των τεστ με ADN ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πρέπει οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε περισσότερες ε, μορφές ελέγχου, σε περισσότερα τεστ. Δεν πρέπει εμείς να παραπέμπουμε στις κυβερνητικές διαδικασίες ελέγχου, δεν κατηγορώ κάποια κυβέρνηση, αλλά οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν τις συνθήκες σωστού ελέγχου. Υπάρχει λοιπόν εδώ ευθύνη για την Ένωση, γιατί αυτά τα οποία αποφασίζονται δυστυχώς δεν, είναι, δεν μένουν πράγματι, δεν εφαρμόζονται με σωστό τρόπο. Και ε, δεν κρύβεται εδώ ο κίνδυνος στον τομέα της υγιεινής που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Κλάες. Κύριε Κλάς, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είναι φανερό ότι πρόκειται για απάτη και η απάτη πρέπει να τύχει καταστολής. Απλώς το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τη νέα νομοθεσία. Έχουμε το βασικό κανονισμό, έχουμε το δίκαιο για τα τρόφιμα, έχουμε την ε, οδηγία για την ετικετοθεσία Όλα αυτά λοιπόν τα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να ισχύουν, θα πρέπει να την χάνουν εφαρμογή και να γίνεται έλεγχος και θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρώσεις για την παραβίασή τους. Και φυσικά θα πρέπει να είναι τέτοιες οι κυρώσεις ώστε να είναι αποτρεπτικές. Τώρα είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αδικαιοδοσία για την προέλευση του κρέατος. Αυτό είναι γραφειοκρατικό και δύσκολο να εφαρμοστεί αλλά θα πρέπει να έχουμε επαρκείς υπηρεσίες ελέγχου για να ελέγχουν. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να έχουμε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, αλλά απλώς να έχουμε πιο στεναρούς και ε, επακριβείς ελέγχους. Έχω ακόμα μισό λεπτό λοιπόν και να σας πω ότι τα βασικά τα έχω πει, οπότε μπορώ να σταματήσω και εδώ. Ο Ζουλ Κανιό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ε, εγκαίρω, προήμως μάλιστα, γιατί πρέπει να πάω στον τριγωνικό διάλογο για τα διαμεθοριακά θέματα. Το σκάνδαλο αυτό μας καταδεικνύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Και λέω σε όλους τους αντιευρωπαϊστές και τους ευρωσκεπτικιστές στο Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, να τους πω ότι αν τα κράτη-μέλη δεν είχαν αρνηθεί να υπάρχει η χνηλασιμότητα και η ε, ετικετοθεσία, δεν θα, στα μεταποιημένα τρόφιμα, δεν θα είχαμε αυτό το σκάνδαλο οποίο μας. Επίσης, πρόκειται και για ένα σκάνδαλο ε, υγειονομικού χαρακτήρα, γιατί στα η φενιλοβουταζόλη που εμφανίστηκε στο αλογίσιο κρέας είναι τοξική για τον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν ένα υγειονομικό πρόβλημα. Και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κύκλωμα που εμπλέκει διάφορες χώρες, ιδίως στη Ρουμανία για τα άλογα αυτά και διαπιστώσαμε υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα μικρό ζωικό κεφάλαιο και μετά από μια τροποποίηση των αποφάσεων της Κομισιόν ένα μεγάλο αριθμό των ε, αλόγων στη Ρουμανία πήρε το δρόμο για τα σφαγεία. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτή η τοξική ε, ουσία λόγω της παρουσίας της Ουκρανίας. Thema Herkunftskennzeichnung ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Χόισλινγκ. Υπάρχει ένα βασικό ζήτημα εδώ πέρα. Λέμε πως πρέπει να παρακολουθούμε από πού προέρχεται το κρέας. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά υπάρχει ε, ελπίδα κάποιοι να αλλάξουν την άποψή τους. Σήμερα στη Γερμανία αποφασίστηκε πως ε, θα ζητηθεί να υπάρξει σήμανση και των συστατικών των έτοιμων τροφίμων. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία η Κομισιόν. Ανησυχούν οι καταναλωτές. Και αν κάνουμε τα γνωστά σχέδια δράσης δεν θα γίνει τίποτα και θα είμαστε όλοι αναξιόπιστοι. Επίσης έχουμε το πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λέμε πώ λύνεται με ελέγχους. Διαφορετικές προδιαγραφές δηλαδή που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Τι θα γίνει. Ε, ο κύριο Μπόργκ υποτίθεται πώ θα συντονίζει όλα αυτά. Γιατί είναι γεγονό, είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές. Αλλού δεν υπάρχουν καθόλου ελέγχοι. Αλλού ελάχιστοι. Επίσης, πρέπει να δούμε και το ρίσκο. Εδώ πέρα διατρέχοντας ελάχιστο κίνδυνο μπορεί κάποιος ε, να κερδίσει πάρα πολλά. Αν δεν το εκμεδενήσουμε αυτό, ε, αυτή τη δυνατότητα αυτού του κέρδους, ε, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ. θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, για μια απάτη παρά τις ρυθμίσεις ε, οι οποίες γίνονται σε διάφορες χώρες για να αποκλιμακωθεί το θέμα, ε, το θέμα ε, δεν αποκλιμακώνεται. Ίσως θα πρέπει να αντιδράσουμε με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε. Μπορεί να μην είναι ο ταχύτερος και ο πλέον διαφανής. Και δεν είναι αλήθεια ότι ε, αν τυχόν είχαμε ψηφίσει για τις ρυθμίσεις που είχαν προταθεί σχετικά με την προέλευση των κρεάτων δεν θα είχαμε το πρόβλημα γιατί έτσι κι αλλιώς ε, η απόφασή μας ε, θα ίσχυε από τον επόμενο χρόνο. Το θέμα είναι λοιπόν πότε θα πάρουμε τις αποφάσεις τελικά που πρέπει να πάρουμε. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχαμε το 2000 τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η βασική στρατηγική προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις να έχουν την βασική ευθύνη, τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τις επιχειρήσεις και η Επιτροπή να ελέγχει τις ελεγκτικές δυνατότητες των κρατών μελών. Αυτή ήταν η λογική. Πού βρισκόμαστε σήμερα, μπορείτε να μας πείτε ε, πού μας έχουν οδηγήσει και πού θα μας οδηγήσουν όλες αυτές οι πολυεπίπεδες διαδικασίες ελέγχου. Μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη με τεράστιο αριθμό θέσεων απασχόλησης και με τεράστιο κοινωνικό ρόλο. Ναι, ευχαριστώ. Εδώ πέρα κατά βάση έχουμε δύο σκάνδαλα. Το ένα είναι η λανθασμένη σήμανση και θέλω να μάθω από την Κομισιόν πώς θα βελτιώσετε τους ελέγχους, πώς θα τους κάνετε ενιαίους για να μην ε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα ξανά και να μην ξανασυμβούν σε κάποια κράτη. Θα κάνετε περισσότερους δείγματοληπτικούς ελέγχους για να αυξηθεί ε, η πίεση στους απαταιώνες. Εν τω μεταξύ το τεστ DNA κοστίζει 20 έως 60 ευρώ. Ε, είναι βεβαίω ε, αρκετά ακριβό για να γίνεται σε καθημερινή βάση. Τι θα κάνετε. Δεύτερον, το δεύτερο σκάνδαλο, η Λουταζόνη, η οποία βρέθηκε μεταξύ άλλων ε, ουσιών, η οποία είναι φαρμακευτική ουσία. Τι θα κάνετε επίσης με το διαβατήριο το λεγόμενο των ε, αλόγων. Θα υπάρξουν εξίσου αυστηροί έλεγχοι για την ειχνηλασιμότητα των ε, νεκρών αλόγων όπως γίνεται με τα βοηδή. Γιατί στα βοηθοί πρέπει να ξέρουμε και τι έγινε το νεκρό ζώο και τα λοιπά, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ, Γιούντιθ Μέρκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το κρέας, ε, ό,τι φαίνεται, των αλόγων ε, πέρασε κάπως και από την Ολλανδία. Οπότε το ζήτημα τι είναι, ότι δεν έχουμε καλούς κανόνες ή επαρκείς ελέγχους. Γιατί ε, βλέπουμε, ε, όπως ε, και με τα αυτοκίνητα και τον κύκλο δοκιμών, βλέπουμε πως βασιζόμαστε σε εθνικές προδιαγραφές. Η διαφορά λοιπόν είναι στην ποιότητα, στη συχνότητα, στην αξιοπιστία των ελέγχων και αυτό οφείλεται στα κράτη-μέλη. Εγώ δεν είμαι υπέρ ενός νέου ελεγκτικού οργάνου κτλ. κτλ αλλά βελτίωση της ίδιας οδηγίας. Και θέλω να ακούσω την άποψη της Κομισιόν. Και τέλος το τι ζητάει ο κύριος ε, Σλούτερ. Δηλαδή ε, αυτό το οποίο κάνουμε, το να θέμε συνέχεια φτηνό κρέας είναι ίσως ε, μια αιτία του προβλήματος. Και για να είμαι ειλικρινής, πριν από δύο ημέρες υπήρξε και μια έκθεση του UNEP, του προγράμματος ε, του ΟΗΕ για την ανάγκη ε, παροχής ε, φτηνού κρέατος. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι το σκάνδαλο αυτό με το ήπιο κρέας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Θα πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα από αυτά τα οποία συνέβησαν έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν στο μέλλον. Τρία είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο είναι της απάτης των εις των καταναλωτών. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί. Το δεύτερο είναι η ασφάλεια στον τομέα της υγείας. Περιλαμβάνονται φαρμακευτικές ουσίες κτηνιατρικές, επικίνδυνες για τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις λόγω της κρίσης και για υπηκούς συλλόγους σε χώρες όπως η Ιταλία και δυστυχώς χρειάστηκαν να απαλλαγούν από ε, ένα συγκεκριμένο αριθμό ζώων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες αγαπούν τα άλογα και δεν θέλουν να τα έχουν στα πιάτα τους. Λοιπόν, τίθεται εδώ και το θέμα της ιχνηλασιμότητας, της ετικετοθεσίας και της αύξησης των ελέγχων. Θα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσες τέτοιες περιπτώσεις βρίσκουμε στην Ευρώπη, πού συγκεντρώνονται οι περισσότερες περιπτώσεις. Έχετε κάποιες εκτιμήσεις, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αντί να τρώει κάποιος βοδινό κρέα σήμερα το βράδυ θα συνεχίσει να τρώει ήπιο. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι πριν από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ κύριε Γιανακουδάκη. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην κάνουμε αυτή την κρίση ευκαιρία για ορισμένου να φέρουν άλλα και άσχετα θέματα στην ημερησία διαταξή. Εγώ ανησύχησα για το γεγονός ότι πάρα πολλοί μιλάνε για θέματα ανιχνευσιμότητας, αλλά θα είχε αλλάξει το να υπάρχει ετικέτα προέλευσης. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το κρέας που έρχεται από μια χώρα θα είναι πιο επικίνδυνο από το κρέας μιας άλλης χώρας. Εδώ έχουμε μια απάτη, είναι φανερό την απάτη. Λοιπόν, αντίθετα θα πρέπει να βλέπουμε τις ευθύνε των παραγωγών των τροφίμων και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πώς μπορούν οι αγοραστές αυτού του κρέατος στα σούπερ μάρκετ να είναι πιο υπεύθυνοι σε σχέση με την ποιότητα και την προέλευση του κρέους αυτού. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για όλα αυτά και θα ήθελα η Κομισιόν να εξασφαλίσει όλη την αλυσίδα από τον παραγωγό ως τον καταναλωτή. Αλλά ίσως και η Επιτροπή κρίμα θα πρέπει να επιληφθεί διότι εδώ μπορεί να υπάρχει πράγματι μια απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Η Έλενα Αντωνέσκου έχει το λόγο. vreau uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα επαληθεύσεων, κυρώσεων και μια ευρωπαϊκή ε, λύση. Προφανώς θέλω να μιλήσω σημερινή συζήτηση γιατί μετά από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι υπάρχει σύγχυση εδώ πέρα ε, όταν μιλάμε ειδικά για τη Ρουμανία και για τον ρόλο που είχε η Ρουμανία ή τη θέση που είχε η Ρουμανία στο σκάνδαλο αυτό. Και θεωρώ πως ε, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως ε, οι κατηγορίες αυτές ήταν αβάσιμες και άδικες. Η Κομισιόν πρέπει να το πει αυτό ξεκάθαρα, γιατί τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν ξεκάθαρα. Η σήμανση είχε γίνει πάρα πολύ σωστά στην Ρουμανία και η χνηλασιμότητα υπήρχε. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα λοιπόν. Οι ρουμανικές αρχές ε, ε, εφάρμοσαν ε, σωστά τις διαδικασίες. Οπότε η απάτη ήταν απάτη σήμανσης και αυτή έγινε εκτός ε, Ρουμανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ για τον κλάδο να ε, βρει τους υπεύθυνου. γιατί η αξιοπιστία του κλάδου αυτή τη στιγμή διακυβεύεται. Σας ευχαριστώ Ρενάτε Ζόμερ. Ευχαριστώ. Ναι, είναι μια απάτη και ε, καμία σήμανση δεν βοηθάει απέναντι στην απάτη. Είχαμε κάνει τον σχετικό κανονισμό και εντός του Κοινοβουλίου υπήρχε μια πλειοψηφία που ήθελε την ε, σήμανση της προέλευσης. Ε, τα κράτη-μέλη δεν το ήθελαν και εγώ είμαι επιφυλακτική για το εάν είναι εφικτό. Γιατί η πλειοψηφία πετούσε σήμανση σε τρία επίπεδα. Δηλαδή τόπος γέννησης, ε, σφαγής και αν επρόκειτο και για επεξεργασμένο κρέας και επεξεργασίας. Και ε, ζητήσαμε από την Κομισιόν να το εξετάσει και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή το εξετάζει σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια σήμανση της ε, προέλευσης και μιλάμε βεβαίως και για το κρέας ε, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία και είναι μέσα σε ολοκληρωμένα προϊόντα. Κάτι θα μας υποβάλει λοιπόν η Κομισιόν μέχρι το τέλος του έτους και να κάνει μια νομοθετική πρόταση. Το ερώτημα λοιπόν προς την Κομισιόν είναι πόσο έχει προχωρήσει. Τέλος, ε, μην αντιδράμε σπασμωδικά και να αποφασίσουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι εφικτό πρακτικά. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μη ρεαλιστικούς νόμους. Και άρα, ε, επίσης, για ένα εθνικό πρόβλημα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πίνες. Πρέπει να κοστίζει ακριβά να κάνει κανείς κάτι τέτοιο και να δημοσιοποιήσουμε το όνομα της επιχείρησης. Ευχαριστώ, Παύλ Πόκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θα επαναλάβω τι τις καλές ιδέες των συναδέλφων. Ε, νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με το σύστημα των γρήγορων ειδοποιήσεων για τα τρόφιμα και τις οτροφές. Μπορούμε να ανταλλάσσουμε μέσω αυτού του συστήματος ε, και πληροφορίες για τις περιπτώσεις τέτοια απάτης. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Μπατ Στάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, σήμανση της προέλευσης. Πράγματι, στο τέλος του έτους η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Κατάλαβα καλά πως συμφωνείτε ε, με το αίτημα των Υπουργών Γεωργίας ε, να κάνετε κάτι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι στο τέλος του έτους. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Μετά, πράγματι είναι μια απάτη εις βάρος του καταναλωτή και πράγματι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να οργανώσουν το σύστημά τους για να είναι σωστή η έλεγχη, να εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και εκεί πέρα φαίνεται πως ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Η Κάρτη Καλλιόρτα ανέφερε το κομμάτι της Ολλανδίας, ε, δηλαδή ο έμπορος που έβαλε λάθος ε, ετικέτα και είχε καταδικαστεί ήδη για το ίδιο πράγμα. Για την ίδια ακριβώς απάτη. Έπρεπε να τον προσέχει το Ολλανδικό κράτος και να κάνει μια ανάλυση κινδύνου. Επίσης, το ερώτημα είναι, όταν κάνουμε ελέγχους, τι κάνουμε μετά. Έχουμε την υπηρεσία ασφάλεια τροφίμων στην Ιρλανδία, κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι 90 άνθρωποι. Τι να κάνουν. Θα πρέπει να ε, και βλέπετε με τον νέο προπολογισμό θα μειωθεί και κατά 5% ο προπολογισμό και το προσωπικό. Απαράδεκτο αυτό. Πρέπει να κάνουμε κάθε χρονιά μία συζήτηση. Τι έχει γίνει, ποιε είναι οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Και από την άλλη είναι και δουλειά των κρατών μελών ο καθένας στη χώρα του να κάνει μια συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να δει τι γίνεται με τις εκθέσεις για την κάθε χώρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Η Βίκη Φόρντ. Ευχαριστώ. Τρία σημεία. Ναι, είναι απάτη, πρέπει να υπάρξει ε, δίωξη και οι πιο αυστηρές πίνες. Χρειαζόμαστε ανιχνευσιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων για να αποφύγουμε την ε, διάδοση ασθενειών. Αν πάμε πίσω στο παρελθόν, είχαν έρθει νεκρές ε, γαλοπούλες στην ε, περιοχή μου και έχουν μεταφέρει ασθένειες και θα μπορούσαν, παρά το γεγονός ότι ήταν πεθαμένες και νεκρές οι γαλοπούλες, να ετικετοποιηθούν σαν βρετανικού χαρακτήρα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα στοιχεία για την προέλευση των τροφίμων. Και ένα επόμενο σημείο, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουμε την αύξηση του πληθυσμού. Αφήστε με να μιλήσω, αφήστε με πώς θα θρέψουμε τον πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται διεκώς. Λένε ορισμένοι δεν θα πρέπει ο κόσμο να αγοράζει φθηνά τρόφιμα, μα δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα άλλο. Ούτε τρόφιμα γενικά δεν μπορούν να αγοράσουν πάρα πολύ. Αγωνίζονται για να τα καταφέρουν. Αν δούμε και σε άλλες επιτροπές ποιο είναι το ποιο, ποιος είναι ο προπολογισμό για την έρευνα στα τρόφιμα. Οι συνάδελφοι αποφασίσανε και δεχτήκανε να περικόψουν εκατομμύρια από τον προπολογισμό για την έρευνα στα τρόφιμα όταν ακριβώς οι καταναλωτές χρειάζονται πιο πολύ έρευνα. Λοιπόν, θυμηθείτε το αυτό το πράγμα και κάντε κάτι. Τέλος, η Σοφία Κονή, η οποία είναι και αυτή η συγγήτρια για το θέμα της ετικετοθεσίας στα ζωικά προϊόντα, στα, στα κρέατα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια απάτη. Ένα έγκλημα, μια εγκληματική ενέργεια. Όπως είπανε πολλοί από τους συναδέλφους, δεν πρέπει να νομοθετήσουμε υπό το κράτος των συγκινήσεων και να μην δώσουμε μια νομοθετική απάντηση σε ένα εγκληματικό γεγονός. Ας δούμε τι έγινε. Καταρχήν, η έρευνα έγινε από την Ευρωπόλ και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει, δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια κάποια αμεροληψία γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομία που κάνει αυτή την έρευνα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν υπάρχουν τέτοιες υποψίες απάτης ζητάμε να είναι η η οποία κάνει την έρευνα γιατί εγώ θυμάμαι την ε, περίπτωση των ε, ε, σπόρων που είχαν έρθει από την Αίγυπτο στη Γερμανία και οδήγησαν σε θανάτους και τότε είχαν κατηγορηθεί οι Ισπανικές αρχές. Λοιπόν, το να γίνεται η έρευνα από την Ευρωπόλ επιτρέπει μια ε, ουδετερότητα και αμεροληψία που εμείς την υποστηρίζουμε. Δεύτερον, το θέμα της πορείας των τροφίμων αυτών δεν οφείλεται στα κρέατα τα ίδια. Πήγανε από τη Ρουμανία στην Νότια Γαλλία όπου κόπηκαν σε κομμάτια και μετά πήγανε στη μεταποίηση. Το θέμα είναι ότι μπορέσαμε να βρούμε μέσα σε λίγες ώρες όλη την πορεία του κρέτος. Το πρόβλημα είναι το θέμα του ελέγχου ή κυρώσει και εκεί πρέπει να είμαστε στεναροί, εκεί πρέπει να είμαστε ικανοί. Τελευταίο ερώτημα, η ασφάλεια των προϊόντων που πρόχονται από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα βρούμε εκεί πέρα για προϊόντα ορισμένων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει ο Σας ευχαριστώ για το 1,5 λεπτό σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Πάολα Τεστόρη ως ε, διευθύντρια, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, αν ξεχάσω κάποια συγγνώμη γιατί τέθηκαν πάρα πολλέ σε πέντε τμήματα η παρουσίαση. Πρώτον, ανιχνευσιμότητα, ηχνηλασιμότητα και νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε πολύ αναπτυγμένη νομοθετική ρύθμιση, την πιο αναπτυγμένη στον κόσμο και χάρη ακριβώ την ρύθμιση αυτή η χνηλασιμότητα είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει. Μπορέσαμε να εντοπίσουμε εμείς την, ε, την αλυσίδα, αν θέλετε, ε, διανομής των προϊόντων μέσα σε λίγες μέρες. Ήταν πιο δύσκολο να βρει κανείς από πού ήρθε το, το πρώτο προϊόν, το βασικό προϊόν. Αλλά είναι δύσκολο να μην αποκαλυφθεί η απάτη. Πάντως παρόλα αυτά από τη Ρουμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο η αλυσίδα αυτή εντοπίστηκε μέσα σε μία ή δύο μέρες και αυτό έγινε ακριβώς χάρη στο σύστημα ανιχνευσιμότητας. Είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που έχουμε αυτή την δυνατότητα που λειτουργεί τόσο καλά. Πριν ζητήσουμε λοιπόν περισσότερη ε, ε, ίχνηλασιμότητα και περισσότερες ρυθμίσεις σε επίπεδο ετικέτας θα πρέπει να το σκεφτούμε. Οι νομικές ρυθμίσεις υπάρχουν. Δεύτερο θέμα, το θέμα προέλευσης. Ακόμα και αν γνωρίζουμε την ε, προέλευση, και δεν θέλω, θέλω να παροθέσει εγώ ε, να, να παροθέσει γύρω στο αν θα πρέπει να υπάρχει προέλευση ε, του κρέατος ως συστατικού σε ε, προπαρασκευασμένα γεύματα. Αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας έκθεσης και του Κοινοβουλίου. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πώς ακριβώς πρέπει να προχωρήσουμε εδώ, τι κόστος θα υπάρχει, εμείς θα προσπαθήσουμε να πάμε πιο γρήγορα, επιταχύνουμε τη διαδικασία, γιατί ο σύνομοθέτης μας ζήτησε να τελειώσουμε την έκθεση αυτή στο τέλος του χρόνου, θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε το φθινόπωρο, αλλά επειδή πρέπει να είναι σοβαρή η μελέτη μας, δεν θα γίνει πριν από το καλοκαίρι όπως το ζήτησαν ορισμένοι υπουργοί. Λοιπόν, το φθινόπωρο όσο πιο νωρίς ε, μπορούμε. Ακόμα και αν η προέλευση θα ήταν υποχρεωτική, η απάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είχε συμβεί. Έτσι και αλλιώ γιατί επρόκειτο περί απάτης ε, και η απάτη αφορούσε το όνομα του είδους, όχι την προέλευση. Υπάρχει απάτη στο συγκεκριμένο είδος του ζώου με λίγα λόγια. Λοιπόν, τώρα μιλώντας πάλι για την απάτη, είναι αλήθεια και το είπαν πολλοί ευρωβουλευτές γιατί δεν επιβάλλεται αυστηρότερες κυρώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ποινικέ κυρώσεις όταν υπάρχουν απάτες στον τομέα των τροφίμων. Κοιτάξτε, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών Κάποιοι ευρωβουλευτές είπαν αν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη. Όχι, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν τις δικές τους εδώ αρμοδιότητες. Οι υπηρεσίες ελέγχου θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις οι οποίες να είναι αποτρεπτικές και σοβαρές, αλλά δεν θα τις πούμε εμείς ποιες είναι. Τώρα, ποιος ελέγχει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Να ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπε η κυρία Μαγκίνες. Κοιτάξτε, αυτό έγινε από έλεγχο της ίδιας της επιχείρησης. Αυτός ο έλεγχος που έκανε η επιχείρηση στα προϊόντα της και βρήκε το κρέας του αλόγου. Και αυτό έγινε γιατί υπήρξε μια επίσημη επιχείρηση, μια επίσημη μορφή ελέγχου στην Ιρλανδία και έτσι η εταιρεία Findus αποφάσισε να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της. Με αφορμή λοιπόν έναν επίσημο δημόσιο έλεγχο σε μία χώρα, μία άλλη επιχείρηση ευτυχώς μπόρεσε να βρει ε, το προϊόν αυτό. Ανακαλύψαμε λοιπόν την απάτη. Η απάτη δυστυχώς είναι ενδογενές χαρακτηριστικό ασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας. Και όπως είπε και ο κύριος Σλούτα, ε, Ξέρετε ότι το ποσοστό των τροφίμων στον οικογενειακό προϋπολογισμό συνεχίζει να μειώνεται. Πριν 15 χρόνια ήταν το 30% του προϋπολογισμού, τώρα είναι 15%. Σε ορισμένες χώρες είναι ακόμα χαμηλότερο και συνεχίζει να κατεβαίνει. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι έμποροι και οι επιχειρηματίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καταναλωτών για χαμηλές τιμές, γιατί οι τιμές είναι η βασική ανησυχία των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης. Χρειάζεται λοιπόν να μπορεί κανείς να κάνει αυτά τα οποία επιτρέπει η εσωτερική αγορά, να αναζητεί δηλαδή τον προμηθευτή στην χώρα όπου είναι ευθυνότερος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η παραγωγή των τροφίμων στην Ευρώπη. Χάρη λοιπόν στην εσωτερική αγορά μπορούμε να πούμε ότι οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν στις χώρες μέλη είναι οι ίδιοι σε όλες τις χώρες πριν σε εισαγωγικά ποινικοποιήσουμε το σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Μιλάμε για συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς, κανόνες ίσοι για όλους που επιτρέπουν στην βιομηχανία των τροφίμων να αναζητά τρόπους ε, ε, μείωσης της τιμής του προϊόντος. Ποια ήταν η ανταπόκριση της Ένωσης. Μέσα σε λίγα λόγια ενημερώθηκαν όλα τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, αν και ασχολείται κυρίως με θέματα υγείας, αλλά εκεί όπου υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει πρόβλημα υγείας και παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας λειτουργήσε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μπορέσαμε να διανύμουμε τις πληροφορίες που είχαμε συλλέξει, να ενημερώσουμε ακριβώς ποια ήταν και η, ε, αλυσίδα που ακολούθησαν τα έτοιμα αυτά ε, τρόφιμα μετά από πληροφορίες των αρμόδιων γαλλικών αρχών. Ε, έχουμε προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης, ε, αλλά είναι σε επίπεδο σύστασης, γιατί δεν έχουμε τη νομική βάση για να προχωρήσουμε σε μια δεσμευτική πρόταση. Είναι μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη, θα την έχουμε έτοιμη αύριο και θα εφαρμοστεί de facto θα χρηματοδοτήσουμε το 75%. Τα τεστ DNA χρηματοδοτούν, ε, κοστίζουν 400 ευρώ κατά περίπτωση και θα χρηματοδοτήσουμε το 75%. Θέλουμε μέσα σε ένα μήνα να έχουμε κλείσει την προσπάθεια γιατί θέλουμε να μην καθυστερήσουμε για μήνες. Θα υπάρξει επίσης και έλεγχος για την φενηλική μπουταζόνη. Γιατί αυτό, γιατί προ στιγμή είδαμε ότι όλα τα ευρήματα οδηγούν στην στρεβλή ετικετοθεσία, στις α, α, απατηλές ετικέτες δηλαδή, αλλά ε, βλέπουμε ότι την ουσία αυτή την είχαν και στο παρελθόν ε, τα δείγματα από ε, κρέας αλόγου. Συνεπώς ο έλεγχος λοιπόν σύμφωνα με την παραγωγή σε κάθε κράτος μέλος είναι κάτι το υποχρεωτικό για την νομοθετική μας ρύθμιση. Και αυξάνουμε τα τεστ αυτά για να διαβεβαιώσουμε τους καταναλωτές και για την ασφάλεια των προϊόντων και να μην σταθούμε μόνο στο είδος του ζώου αλλά και στην ασφάλεια της κατανάλωσής του. Τώρα κάποιες άλλες παρατηρήσεις, ερωτήσεις για την κλωνοποίηση. Κοιτάξτε, για την κλωνοποίηση. Εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να παραμείνουμε στην μελέτη της, ε, ε, της, των επιπτώσεων. We will make a my took the to make a Την αξιολόγηση της, των επιπτώσεων της ρύθμισης αυτής και στα πλαίσια του κανονισμού για την υγεία. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να καταστήσουμε τους κανονισμούς για την υγιεινή και υγεία πιο χαλαρούς. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές που είναι η ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση των εθνικών αρχών. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνε για τον έλεγχο των σφαγίων και των επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος. Αλλά παρόλα αυτά ε, κάποιες ε, ε, διαδικασίες επιτρέπεται να γίνουν από ορισμένε επιχειρήσεις όπως η δειγματοληψία. Αυτό ισχύει στα κοτόπουλα σαν παράδειγμα. Και θα πρέπει ο έλεγχος αυτός να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κινδύνου κάθε φορά. Δεν προτείνουμε αλλαγές δηλαδή ριζικές, αλλά μία πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες και μία μεγαλύτερη ε, ε μείωση ε, της γραφειοκρατίας, γιατί ένα τμήμα του Κοινοβουλίου ζητάει περισσότερες νομικές ρυθμίσεις και ένα άλλο τμήμα του Κοινοβουλίου ζητάει συστηματικά λιγότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Τι αποφάσισαν οι υπουργοί την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αποφάσισαν τίποτα. Στο θέμα αυτό θα είναι στη μέση διατάξη γιατί είναι γεγονό ότι υπήρξε μεγάλη πολιτική ανησυχία. Δεν ελήφθη όμω καμία απόφαση. Θα υπάρξει και πάλι αίτηση προ την Κομισιόν να προχωρήσει πιο γρήγορα στην τυχετοθεσία προσέλευση. Γιατί η διακατάσταση που αντιμετωπίζουμε στο Κοινοβούλιο, οι μισοί θέλουν περισσότερη ετικετοθεσία και οι άλλοι λιγότεροι, γίνεται το ίδιο πράγμα και στο Συμβούλιο. Πόσους ελέγχους ε, διενεργούμε στον τομέα των τροφίμων, είμαστε τυχεροί. Γιατί είναι ο μόνος τομέας πολιτικής μαζί με την πυρηνική ασφάλεια και με την αλληλεία που να έχει ανεξάρτητο σώμα επιθεωρητών που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τομέα του περιβάλλοντος δεν έχετε. Στα τρόφιμα έχουμε 110 ελεγκτές που επιτηρούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι από τα κράτη-μέλη. Κάνουν 200 με 300 ε, επιθεωρήσεις στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτών δημοσιεύονται. Χάρη σε αυτούς τους ελεγκτές μπορούμε να πούμε ότι η τροφιμική μας αλυσίδα είναι ασφαλής, ότι είναι υγιής δεν πρέπει να θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στην τροφιμική μας αλυσίδα. Υπάρχουν περιπτώσεις απάτης και πάντα θα υπάρχουν απάτες, αλλά είναι πολύ περιορισμένες. Προσπάθησα κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον προσπάθησα να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δεστόρη και έχουμε και την Εύσα εδώ πέρα σήμερα. Βεβαίω θέλουμε να την ακούσουμε. Ο κύριος Μπερνάρ, Διευθυντής Αξιολόγησης ε, Κινδύνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ που μας δίνετε και εμάς την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ήδη η κυρία Τιστόρη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, κίνδυνος ε, για την ασφάλεια τροφίμων είναι ένα ζήτημα απάτης και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας τροφίμων και η ΕΦΣΑ πέρα από τα κατάλοιπα των τροφίμων βοηθάει και αυτούς που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνου ε, και στην περίπτωση αυτή γιατί τώρα με βάση την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργαζόμαστε για τον εξυγχρονισμό του συστήματος επιθεώρησης του κρέατος. Ε, η σύστασή μας θα βγει τον Ιούνιο. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση αυτή, υπάρχουν μόνο τρεις ε, τομείς ανησυχίας. Ε, το ένα είναι ένα παράσιτο της τριχινίασης που είναι πάρα πολύ σπάνιο αλλά μπορούν να προσβληθούν από τριχινίαση και τα άλογα, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο ένα στα 100.000 άλογα, οπότε δεν είναι μεγάλη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, αλλά ε, υπάρχει μια πιθανότητα. Τώρα, για τα φαρμακευτικά, το ένα είναι η φετοβεναζόλη που ήδη αναφέρθηκε, που είναι αντιφλεγμονώδες, που χρησιμοποιείται και στους ανθρώπους ε, για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, ε, αρθρίτιδας στους ανθρώπους και χρησιμοποιείται και στα άλογα υποδρόμου, αλλά είναι σαφές πως τα άλογα αυτά δεν επιτρέπεται μετά να μπουν στην τροφική αλυσίδα. Ε, αν γίνει κάτι τέτοιο βεβαίως είναι ένα λάθος ε, στην ε, διατροφική αλυσίδα, αλλά υπάρχουν οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έχουν ελεγχθεί χιλιάδες δείγματα τα τελευταία χρόνια και ε, ελάχιστα από αυτά ε, δείχνουν αυτή την ουσία. Και τέλος θα έλεγα πως ε, ε, ως χημικό κατάλοιπο έχουμε κάδμιο στο κρέας των αλόγων, αλλά και πάλι είναι Ελάχιστο κίνδυνο, απλά ανοιχνεύεται γιατί το αναζητούμε. Οπότε θα έλεγα συνολικά πως το κρέας των αλόγων και από πλευρά μικροβιολογικής είναι πολύ ασφαλές. Οπότε και ομό μπορεί να το φάει κανείς χωρίς ε, κίνδυνο. Ε, το θέμα της απάτης είναι, ε, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν είναι ζήτημα ε, υγιεινής. Και βέβαια η ΕΦΣΑ είναι στη διάθεσή σας ε, με τα νέα δεδομένα για να βοηθήσει, γιατί τώρα βεβαίως θα ενταθούν οι έλεγχοι και συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων για να βοηθήσουμε αυτούς που κάνουν τον αξιολόγηση του κινδύνου για να επαναξια... επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει η συζήτηση. Ο Κρις Ντέβις ένα συμπληρωματικό ερώτημα ήθελα να θέσει. Αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρο. Αν θα επιτρέψετε κάποια συμπληρωματικά ερωτήματα ή τουλάχιστον ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Κυρία Τεστόρη, πρέπει να φύγετε σε πέντε λεφτά. Πάρα πολύ σύντομες ερωτήσεις λοιπόν. Η Λίνα Μακιέβεν και ο Κρυς Ντέβις. Εντάχει παρακαλώ. Μαγκίνες, συγγνώμη. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ένα μονάχα. Λίντα. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τεστόρη. Το να έχουμε ετικετοθεσία στα ζωικά προϊόντα. Δεν είναι ο σκοπός οι εταιρείε να έχουν περισσότερη ευθύνη για το τι βάζουν στα προϊόντα. Δεν άκουσα τίποτα από την Κομισιόν σήμερα που να λέει στον καταναλωτή κάτι καθησυχαστικό ότι κάτι θα αλλάξει. Ναι, έχουμε ένα σύστημα. Ένα σύστημα που απέτυχε. Δεν ήταν μία εταιρεία, πολλές εταιρείε. Μιλήσατε για γραφειοκρατία. Μα πόσα θα δαπαρίσουμε τώρα για τις δοκιμασίες για να προσπαθήσουμε να αναπτερώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αν δεν θέλετε την ετικεφεσία για τα, ζωικά, για τα προϊόντα κρέατος, με ποιο τρόπο θα υπευθονοποιήσετε τις εταιρείες για να ξέρουν από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά. Ο εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι είναι οι καλύτεροι νόμοι στον κόσμο, οι νόμοι περί ετικετοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και από τι εθνικέ κυβερνήσει. Αλλά βλέποντα την νομοθεσία, δεν βλέπω πώ οι εθνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή τη ρήτρα. Είναι 27 διαφορετικέ μέθοδοι που ακολουθούνται. Δεν ξέρω ότι δεν είναι μονάχα αυτό για τα τρόφιμα, είναι και για πολλά άλλα προϊόντα μπορεί μερικά κράτη να ελέγχουν, άλλα να μην ελέγχουν. Δεν έχουμε καθόλου στοιχεία δεν έχουμε κάποια συλλογή στοιχείων που να δείχνει πώ γίνεται η επιβολή τη νομοθεσία και ποιε είναι οι κυρώσει που επιβάλλονται σε περιπτώσει παραβιάσεων. Μαγκίνε. Σα ευχαριστώ. Το δικό μου ερώτημα άπτεται τη ΕΦΣΑ και τη σχέση τη με άλλου φορεί όπω είναι ο φορέα τροφιμική ασφάλεια στην Ιρλανδία. Ξέρω ότι ο κάθε φορέα έχει διαφορετικέ αρμοδιότητε επί τη βάση του τι του επιτρέπουν οι εθνικέ αρχέ. Και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν πόσο δύσκολο να είναι συνεκτικέ όλε αυτέ οι διαδικασίε. Η Ιρλανδία εξέταζε την αυθεντικότητα των τροφίμων, γιατί το αποφάσισε αυτό η ίδια η Υπηρεσία Τροφιμική ασφάλεια στην Ιρλανδία, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γίνεται. Αλλά εγώ ε, αναρωτιέμαι αν έχουν πράγματι την ίδια εντολή και αρμοδιότητα οι φορεί στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε στον Πρεσβευτή ότι αφαίρει η αρμοδιότητα των φορέων στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας για να έχουμε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα στο τι κάνουν αυτοί οι φορείς και να μπορούμε να σεβαστούμε ότι υπάρχει πράγματι ανεξαρτησία, είναι δηλαδή διαθέσιμη πληροφορία στον καταναλωτή μόλις διακριβωθεί. Ναι. Και είναι γεγονός ότι συνέχεια βγαίνουν νέες περιπτώσεις, η περίπτωση του Γκούλας, στη Νότια Γερμανία το μολυσμένο κρέας. Είμαστε λοιπόν όλο και περισσότερα θύματα και όχι θύτες και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε το καλύτερο σύστημα μεν, αλλά όταν έχουμε όλο και περισσότερα σκάνδαλα θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αν φτάνει αυτό το επίπεδο ετικετοθεσίας ή αν θα πρέπει να ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές για τα ζωικά προϊόντα. Το 2001 όταν υπήρχε αυτή η ευκαιρία να το κάνουμε, έλεγε το Συμβούλιο ότι όλο θα κάνουμε ε, περισσότερα πράγματα και περισσότερες κυρώσεις και μετά το απέρριψε αυτό το νομοθέτημα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι καλό το σύστημά μας και επομένω δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν, δεν υπάρχει, κάποιο, όταν υπάρχει κάποια απάτη. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει 100% ε, ασφάλεια, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας τι γίνεται. Έχω πάρει άπειρες ερωτήσεις για το θέμα αυτό και υπάρχει πραγματικά έλλειψη εμπιστοσύνης στην ασφάλεια του συστήματος. Ναι, δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά, αλλά όταν ο καταναλωτής σχεδόν σε κάθε σούπερ μάρκετ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει, ε, παίρνει αλογίσιο κρέας αντί για βόηο κρέας, δεν μπορούμε να κρατάμε τα χέρια μας ψηλά και να μην κάνουμε τίποτα. Κυρία Τεστόρη. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι τόνοι οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την απάτη ήταν γύρω στους 20 τόνους. Αυτό γνωρίζουμε. 20 τόνοι από 100.000 περίπου που καταναλώνονται στην Ευρώπη. Αναφέρομαι σε κρέας από άλογα. 0.02 of the horse meat which circulates in Europe. Δηλαδή το 0,2% του κρέατος αυτού του είδους. Κοιτάξτε, είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι μία πάτη. Μία πάτη είναι σοβαρή. Αλλά ας πούμε στον καταναλωτή μας, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας, Κοιτάξτε, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 2.250 ε, ελέγχους που κοστίζουν όπως είπε ο καθένας 400 ευρώ γιατί θέλουμε να δούμε ποια είναι η διάσταση του προβλήματος. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μεγαλύτερη η απάτη, έχετε δίκιο ίσως πρόεδρε, αλλά προς το παρόν είμαστε σε αυτό που σας είπα. Μία απάτη πολύ σοβαρή, μεγάλη απάτη γιατί αφορά 20 τόνους, αλλά δεν μιλάμε για ένα σύνολο σύστημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο εμείς λέμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε για ένα μήνα να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις μορφές ελέγχου έτσι ώστε να γνωρίσουμε το ταχύτερο δυνατόν την κατάσταση με το ήπιο κρέας στην Ευρώπη. Λοιπόν, τον Απρίλιο θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Σε αυτή τη φάση αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το σύστημα ελέγχων μας και το σύστημα ειχνηλασίας μας δουλεύει, δούλεψε, δουλεύει. Το θέμα της, ετι... της προέλευσης στις ετικέτες είναι κάτι το οποίο θα πιέσει ε, τους ε, επιχειρηματίες να μην χρησιμοποιούν μερικές φορές ε, τις επιχειρήσεις να μην αγοράζουν από άλλες χώρες κρέας. Οπότε τι θα κάνετε, θα επανεθνικοποιήσετε την εσωτερική αγορά. Αυτό είπατε. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση ε, με το τι συμβαίνει με τις υπηρεσίες ελέγχου στις διάφορες χώρες. Σε ορισμένες χώρες ε, ο έλεγχος γίνεται από τα Υπουργεία. Σε άλλες περιπτώσεις ο έλεγχος γίνεται από τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, όπως το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έλεγχος γίνεται από τους δικούς μας επιθεωρητές. Γιατί σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κοιτάξτε, άμεση σχέση ε, και κάθε χώρα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, άλλες μέσω υπουργείων και άλλες μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Εγώ δεν θα προτείνω ένα ενιαίο μοντέλο, εγώ δεν θέλω να θίξω την ελευθερία των κρατών μελών να οργανώσουν τις δικές τους υπηρεσίες. Αυτό που έχει σημασία είναι οι ε, συμβουλές οι επιστημονικές να είναι ανεξάρτητες και διαφανείς και να είναι εξίσου ισχυρές οι μορφές ελέγχου τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να έχουν ελεγκτές και οι ελεγκτές θα πρέπει να ε, μας δείχνουν ακριβώς πώς θα πρέπει να κάνουν αυτές, να αποδεικνύουν πώς κάνουν αυτές, ε, αυτούς τους ελέγχους. I think that Linda want to answer. <laughs> Linda möchte kurz das klarstellen, weil das hat... Η κυρία Μακέβαν ήθελε να κάνει μια διευκρίνηση. Πάολα, όχι, δεν λέω ότι ο στόχος της ετικετοθεσίας είναι να μην μπορούν να κάνουν εισαγωγές κρέατος από άλλες χώρες. Απλώς να ζητήσουμε από τις εταιρείε να κάνουν την ετικετοθεσία για να ξέρουν οι ίδιες από πού έρχεται το κρέας. Οπότε η Φίντους όταν κάνει λαζάνια θα πρέπει να ξέρει όλη την αλυσίδα παραγωγής. Και τότε θα φροντίσει περισσότερο τα λαζάνια της. Όλα αυτά που είπες αφορούν κόστος που τελικά το επομίζεται ο φορολογούμενος. Λέτε ότι τα κράτη, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν κάνει περισσότερο έλεγχο σε μια εποχή λιτότητος και αυστηρότητος. Μήπως υπάρχει και μια πρόταση από την Κομισιόν ώστε οι εταιρείε να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ε, τροφιμική αλυσίδα. Πώς θα πείσουμε τις μεγάλες εταιρείε να αναλάβουν ευθύνη για τα προϊόντα που πουλάνε στο ευρύ κοινό. Ωραία. Μετά από αυτήν την ε, διευκρίνηση η κυρία Τεστόρη έχει την ευκαιρία να απαντήσει εφόσον το επιθυμεί και θα κλείσουμε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο έλεγχος θα πρέπει να παραμείνει τελικά στις αρμόδιες αρχές. Πρέπει να υπάρχει επίσημος έλεγχος. Και η εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει για τον επίσημο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είναι αυτή είναι τα κράτη-μέλη που πληρώνουν. Εμείς θα, θέλουμε να περάσουμε αυτή την ρήτρα ότι οι εταιρείε θα πρέπει να πληρώνουν το κόστος του επίσημου έλεγχου, αλλά πρέπει να παραμείνει ο επίσημος έλεγχος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει στο πέρας της συζήτησης. Πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η συζήτηση αυτού του θέματος. Νομίζω ότι πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από αυτή τη συζήτηση και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε κάποιο συνάδελφο με την ευκαιρία. Αύριο ψηφίσουμε, θέτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας και σας εύχομαι καλή βραδιά.